Uh, Καλημέρα συνάδελφοι. Καλωσορίσατε στην ε, τακτική συνάντηση Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας αρχίσουμε με 20 λεπτά καθυστέρηση. Οι συντονιστές είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γιατί το θα είναι στην ώρα τους εδώ οι συνάδελφοι. Μπάς περιπτώσει, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, την έχετε στους ε, φακέλους σας έχουν διανομηθεί. Θα ήθελα να σας προτείνω μια αλλαγή. Το σημείο 12 θα συζητηθεί αμέσως μετά το σημείο 9. Πρόκειται για τον εξέτες του σχεδίου πρώτας ψηφίσματος της διαπραγματεύσης με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση-ΥΠΑ. Τώρα, προτείνω να αναβληθεί για αργότερα ε, η συζήτηση του σημείου 8 για την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ο συντάκτης, ο Ρόμπερτ Στέρντι, μου είπε ότι υπάρχουν συμβαστικές τροπολογίες, άρα δεν θα συζητήσουμε αυτές που προβλέποντας. Έχει καλώς. Λοιπόν, επανέρχομαι στη μέρη στη διάταξη, σημείο 2 έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας στις 20-21 Φεβρουαρίου. Ο συνήθως θα θεωρηθούν εγκεκριμένα εάν δεν υπάρξουν, ως έχουν να μην υπάρξουν παρατηρήσεις ως το τέλος της συνεδρίασης. Σημείο 3. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, αν μεταδίδεται από το ίντερνετ τη συνεδρίαση, εκτός της συνεδρίας των συντονιστών που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Σημείο 4. Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής για το έτος 2013. Όπως ξέρετε, το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για φέτος άλλαξε μετά από απόφαση που έλαβε η διάσκεψη των Πρόεδρων τον Ιανουάριο μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εβδομάδα του Στρασβούργου και κατά συνέπεια χρειάστηκε να γίνει για το δεύτερο εξάμεινο κάποιος νέος προγραμματισμός ε, των συνεδριάσεων των επιτροπών μας. Το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει ήδη συζητηθεί και με τους ε, συντονιστές. Τώρα, κοινή συζήτηση των σημείων 5 και 6. Πρόκειται για το ίδιο θέμα. τροποποίηση της απόφασης 2125 και 97836. Πρόκειται για τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση συμφωνιών που αφορούν την, ε, ε, την ίση Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ε, μηχανοκίνητα για τους τεχνικούς κανονισμούς που φορούν τα τροχοφόρα οχήματα. Το 1997 ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση την, ε, τον κανονισμό 1958, την ε, παράλληλη συμφωνία και άλλοι είναι η αναθερμένη συμφωνία του 1958. Όλα αυτά έγιναν για να μπορέσουμε να αναπροσαρμοστούμε σε σχέση με την συνθήκη. και γενικότερα με την εξωτερική εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι συντάκτης και, και των δύο εκθέσεων Υπάρχουν και τροπολογίες που αφορούν αυτές τις εκθέσεις και όλα θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες επιτροπές που ενδεχομένως ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό θα ε, γνωμοδοτήσουν πρόκειται για την Ήτρε, την Ίμκο και την Τραν, τις μεταφορές. Πριν να δώσω το λόγο συναδέλφους για να αρχίσει η συζήτηση, το σχέδιο γνωμοδότησης, θα ήθε, συστάσεων που θα επιβάλλω, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση για την επιτροπολογία. τα θέματα αυτά είναι θέματα τα οποία είχαν εγκριθεί πριν από τη νέα συνθήκη και την διαδικασία της επιτροπολογίας την πρώτερη. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει και τις νέες τροπολογίες που αφορούν αυτά τα δύο θέματα. Το σχέδιο συστάσεων το έχετε. Θα ήθελα να πω ότι ακόμη το Συμβούλιο δεν μας έχει ζητήσει να γνωμοδοτήσουμε. Προκαταβάλουμε λοιπόν, προκαταλαμβάνουμε λοιπόν μια κατάσταση. Τον Απρίλιο θα μας ζητηθεί. Να επιληφθούμε του θέματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε αυτό το θέμα. Ο κύριος Δεκάσπερη από το ΕΛΚΑ και με την Καζάλκα, οπότε ε, θέλουν να κάνουν καμία ε, παρατήρηση στα πλαίσια της συζήτησης. Οι δύο συνάδελφοι ήταν οι ισχυώδες συγητές που ανέφερα. θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Είναι η τρίτη φορά που συζητείται αυτό το θέμα. Οι φιλελεύθεροι ζήτησαν, οι άλλοι δεν ζήτησαν λόγο. Όχι, όχι. Κυρία συνάδελφος. Όχι, δεν είχα τίποτα να προσθέσω. Ε, εκτός από το να προειδοποιήσω για κάτι. Καλό είναι το ότι έχουμε παγκόσμιες συμφωνίες, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να είναι ευέλικτες, γιατί όπως είδαμε στην Ήτρε, ε, έγιναν πιο αυστηρές οι διαδικασίες δοκιμών των αυτοκινήτων. Πρέπει να είναι λοιπόν αρκετά ευέλικτες συμφωνίες για να μπορούμε να εισαγάγουμε καινοτομίε. γιατί είναι τόσο μεγάλες και μια φορά οι συμφωνίες που αλλάζουν πάρα πολύ αργά. Αλλιώς χαίρομαι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Μάλιστα, ευχαριστώ είναι αρκετά ευέλικτες κατά την άποψή μου. Βεβαίω, οι αποφάσεις είναι στο φάκελό σας. Κανείς δεν έχει ζητήσει να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Α, σας ακούσουμε την Κομισιόν. Έχουμε την κυρία Ρωμάου από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, την τη Μαργαρίτα Ρουμάου. Πού είσαστε? Εκεί, μάλιστα. Ε, thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν είναι πολύ χαρούμενη που το Συμβουλίο καλωσορίζει αυτές τις δύο προτάσεις. Όπως είπατε ήδη, είναι πολύ σημαντικές. Λόγω της διάστασης ε, των κανονισμών που υιοθέτηθηκαν τα τελευταία χρόνια ε, στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία βασίζεται όλο και περισσότερα σε αυτούς τους κανονισμούς, που φυσικά αποτελούν το αντικείμενο ενδελφούς διαπραγμάτευσης από την Κομισιόν στη Γενέβη. Για να απαντήσω στο σχόλιο που ακούσαμε, ελπίζουμε ότι το σύστημα θα είναι αρκετά ευέλικτο και έτσι θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές, τεχνολογικές εξελίξεις. Έχουμε διαρκώς τροπολογίες για τους υπάρχοντες κανονισμούς που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Όσον αφορά τις διατάξεις ΠΡΑΚ, πράγματι αυτή η νομοθεσία όπως και όλες οι άλλες πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ουσιαστικά αυτό είναι ένας από τους σκοπούς αυτής της άσκησης. Όλες οι αναφορές ε, ΠΡΑΚ που παραμένουν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής ε, να διορθωθούν. Και τώρα στην ε, τελευταία έκδοση που θα στείλει επίσημα το Συμβούλιο θα έχουν μεριμνήσει και για αυτό. Ευχαριστώ. Thank you uh, we have not yet been brief... ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα για την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Αναμένουμε το Συμβούλιο. Βεβαίως υπάρχει περιθώριο για να υποβληθούν τροπολογίες. Είναι κάπως απλή η διαδικασία. Σημείο 7. εμπόριο πρόδρομων ουσιών μεταξύ της κοινότητας και τρίτων χώρων. Το έχουμε συζητήσει τουλάχιστον δύο φορές. Έχουμε συζητήσει το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Προύστ από το ΕΛΚ και τις εννέα τροπολογίες. Ας τις δούμε και ας δώσουμε τον λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όσες και όσους ε, συμμετείχαν στο σχέδιο έκθεσής μου. Θα είμαι πολύ σύντομος, επειδή όπως είπατε έχουμε ήδη συζητήσει πολύ για αυτή την έκθεση και για τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Όπως είπατε, έχουν υποβληθεί εννέα τροπολογίες. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμούς ε, για τις περισσότερες. Αφορούν την ενσωμάτωση των φαρμάκων στις διαφαθμισμένες ουσίες ε, και ειδικότερα τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και τέλος αφορούν την επιτροπολογία. Θα κάνω πολύ γρήγορα προτάσεις ε, συμβιβασμών και για τους κοιόδες συζητητές. Θα ήθελα να επιφοληθούμε αυτή τη συζήτηση για να μελετήσουμε το ενδεχόμενο να λάβουμε μια εντολή από την ε, Επιτροπή Ίντα να προχωρήσουμε σε τριμερή διάλογο ώστε να επιτύχουμε μια ανάγνωση πρώτη, μια ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Η κατάσταση είναι ανησυχητική όσον αφορά την κυκλοφορία φαρμάκων που περιέχουν εφεδρίνη και ψευδοεφεδρίνη. Είναι λοιπόν επίγοντο το ζήτημα και πιστεύω ότι η ποιότητα αυτή τη έκθεση βασίζεται στο πόσο γρήγορα ε, παρέχει δυνατότητες αντίδραση. Πρέπει λοιπόν να παρέχουμε μια απάντηση το συντομότερο δυνατόν. Οι συζητήσει του Συμβούλου έχουν προχωρήσει γρήγορα, η Ιρλανδική Προεδρία δείχνει ιδιαίτερη βούληση για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σα και εννοείται ότι παραμένω ανοιχτός στις προτάσει σα και ανυπομονώ να ακούσω τα διάφορα σχόλιά σα. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τους κοιόδες. Κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής που θα ήθελε να παρέμβει. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος το λόγο. Ας ακούσουμε την Κομισιόν. Που βρίσκεται... Ποιος βρίσκεται εδώ εκ μέρους της Κομισιόν. Θα μπορούσατε να μας πείτε το όνομά σας για τα πρακτικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που υπέβαλαν τροπολογίες για να βελτιωθεί το κείμενο της Κομισιόν. Επίσης, χαιρόμαστε για το ότι ο εισηγητής ε, θέλει να προχωρήσει σε τριμερή διάλογο μόλις εγκριθεί η έκθεση στην Επιτροπή. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Βιέννη εκπροσωπώντας ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα των ε, ναρκωτικών και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ε, νομοθεσία μας, οπότε σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο μόλις η Επιτροπή σας υιοθετήσει το σχέδιο έκθεσης. Για τα ζητήματα αυτά όσον αφορά την ε, προστασία των ε, δεδομένων θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεργαστείτε στενά και με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που επίσης ε, προετοιμάζει μία έκθεση για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών στην εσωτερική αγορά και αφορά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων για να έχουμε παρόμοιες διατάξεις. Τώρα, για τις προτάσεις. Για τον ορισμό αυτών των ουσιών και τη συμπερίληψη των φαρμάκων σημειώνουμε το ότι υπάρχει θέληση να καλυφθεί αυτός ο ορισμός, αλλά μπορούμε να καθαρίσουμε το ποια φάρμακα εξαιρούνται από τον ορισμό και ποια συμπεριλαμβάνονται, αλλά νομίζω πως είναι απλά ζήτημα διατύπωσης και όταν μιλάμε για την ε, τροπολογία 28 εκεί πέρα προτείνεται να επεκταθεί η διαδικασία έγκρισης για όλες αυτές τις ουσίες εδώ πέρα για Τη ουσία κατηγορία 3. Ε, Οι ουσία κατηγορία 3 είναι λιγότερο επικίνδυνε από αυτές κατηγορία 1. Δεν ξέρουμε γιατί προτείνεται αυτό. Και τέλο όσον αφορά την τροπολογία 29 για την ε, επιτροπολογία και την εκχώρηση εξουσιών βλέπουμε πως ε, το σχέδιο έκθεσης από ό,τι φαίνεται και με τις ε, τροπολογίες δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελε η Κομισιόν τέλος. Για την τροπολογία 30 υπάρχει μια πρόταση που λέει πως η Κομισιόν πρέπει να αξιολογήσει την λειτουργία ε, του κανονισμού μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Δεν φτάνει ο χρόνος γιατί από όταν θα τεθεί ενισχύ ε, είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να αξιολογήσουμε κιόλας. Ευχαριστούμε, Καρολίν ο συγητής, κάποια αντίδραση στις αντιρρήσεις ε, της Κομισιόν. Όχι αυτή τη στιγμή. Ας ε, αναμείνουμε λοιπόν τις συμβαστικές τροπολογίες, εάν υπάρξουν. Θα είναι καλοδεχόμενες. Χρονοδιάγραμμα έγκριση στην Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή μας στις 24 και 25 Απριλίου. Το 8 ακυρώθηκε όπως σας ανακοίνωσα. Because there is no need to... Γιατί δεν θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, γιατί όλες οι συμβαστικές τροπολογίες ε, αποτέλεσαν αντικείμενο συμφωνία με τον Ρόμπερτ Στέρντι, τον εισηγητή. Σημείο 9. Εμπορικές σχέσεις με την Νορβηγία. Εξέταση ερωτήματο ε, με το οποίο ζητά, ζητείτε ε, απάντηση από την Κομισιόν και σχέδιο ψηφίσματος. Τα πράγματα έχουν ω εξή τον Ιανουάριο η ευρωπαϊκή εξαγωγή κάποιων τυριών ε, βορείου κρέατος ε, και αρνήσιου κρέατος αντιμετωπίζουν ε, δασμούς ύψους 277%, 429% και 344% αντιστοίχως. και είχε προηγηθεί δε δασμός εισαγωγικός 72% στις ορτανσίες. Το Νοέμβριο τα είχαμε συζητήσει αυτά τα θέματα με τον ε, Νορβηγό πρέσβη. Οι συντονιστές ε, αποφάσισαν ε, να απευθύνουν μια προφορική ερώτηση στην Κομισιόν και να υποβληθεί και ψήφισμα οι αρμόδιες επιτροπές συμφώνησαν, ξέφρασαν τη στήριξή τους, υπέβαλαν και κάποιες προτάσεις. Οι δε τροπολογίες Επιτροπής θα έρθουν μέσω των πολιτικών ομάδων. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το σχέδιο ψηφίσματος. Για το σχέδιο ψηφίσματος η θα οριστεί μια προθεσμία για τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μα τον Απρίλιο. Ναι. Για την δε ερώτηση δεν θα υποβληθούν τροπολογίε. Οι ομάδε θα τα κάνουν μόνε τους. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Φιέλνερ από το ΕΛΚ που είχε δραστηριοποιηθεί στο θέμα αυτό και τον ευχαριστώ για τον ρόλο του. Κρίστοφερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Πρώτα απ' όλα να πω πως είναι λυπηρό το ότι η πρώτη φορά που μιλάμε για την Νορβηγία στην Επιτροπή μας ε, είναι στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης γιατί η Νορβηγία είναι σημαντικός εταίρος και καλός φίλος μέσω της συμφωνίας ε, για τον ΕΟΧ έχουμε νομίζω μια καλή συνεργασία. Αλλά είναι η πρώτη πραγματική συζήτηση που γίνεται για την Αφρική τα τελευταία νέα χρόνια. Νομίζω πως η Κομισιόν τα είπε ξεκάθαρα στη συνάντηση με τον ε, κύριο Πρέσβη στην Επιτροπή μας όταν είπε πως η Νορβηγία παραβίαζε και το πνεύμα και το γράμμα της ε, συμφωνίας με την εισαγωγή αυτών των ε, δασμών. Καθώς έχουμε δεσμευτεί, σύμφωνα με το άρθρο 19.2, και εμείς και αυτοί, να απελευθερώσουμε το ε, εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Παρά το ότι δεν είναι μέρος επίσημου του πρωτοκόλλου, έχουμε πει πως αναλαμβάνουμε να απελευθερώσουμε το εμπόριο αυτό. Και δεν αντιλαμβάνουμε τι απελευθέρωση είναι αυτή. Δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, πέρα από την νομική πτυχή, ε, δεν τα κάνει κανείς αυτά σε φίλους. Και χωρίς να ε, διαβολευτούν μαζί μας. Ο λόγος ε, για το ερώτημα βέβαια προς την Κομισιόν είναι πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την κλιμάκωση, γιατί δεν είναι προς το συμφέρον ούτε το δικό μας, ούτε της Νορβηγίας, το να αρχίσουμε να αυξάνουμε τους δασμούς. Πρέπει ανταυτού να πείσουμε την Νορβηγία να μην επιβάλλει τους δασμούς και να ε, ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω απελευθέρωση. Για να... και στον τομέα της αλληλείας. Αυτό έχει γίνει επιτυχώς με την Ισλανδία που επίσης είναι στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Μπορεί να γίνει νομίζω και με την Νορβηγία. Τέλος, αντιλαμβάνομαι πως το συζητάνε αυτό το θέμα στην Νορβηγία και βλέπω πως ο ο υπουργό Γεωργία είπε πως δεν θα επηρεαστεί το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Πρώτα απ' όλα το αμφισβητώ αυτό, αλλά ακόμα και αν λέει την αλήθεια, είναι ακόμη πιο περίεργο, γιατί ε, τότε γιατί επιβάλλουν αυτούς τους δασμούς εάν δεν επηρεάζουν το εμπόριο. Γιατί το κάνουν αυτό σε φίλους εάν δεν αναμένουν κάποιο αποτέλεσμα στο ύψος του εμπορίου. Οπότε αναμένω την απάντηση της Κομισιόν και ένα ψήφισμα για να στείλουμε και εμείς το δικό μας μήνυμα για το πώς ε, μπορούμε να αποκλιμακώσουμε αυτή την σύγκρουση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ σε κάποιο βαθμό εκτός από το γεγονός ότι Κρίστοφερ στη δική μας χώρα έχουμε μια ακροδεξιά ομάδα και ένα μέλος κάθε σε αυτή την επιτροπή που υπάρχει σήμερα και που χρησιμοποιεί τη Νορβηγία ως υπόδειγμα μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητείτε ευρέω ότι η Νορβηγία ουσιαστικά λαμβάνει όλα τα ωφέλη χωρί να αντιμετωπίζει κανένα από τα προβλήματα ή τα κόστη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λοιπόν με ανησυχεί ιδιαίτερα. Έχετε δίκιο, είναι φίλοι, έχετε απόλυτο δίκιο στο όσα λέτε. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουμε μια ερώτηση στην Κομισιόν, αλλά η Κομισιόν νομίζω δεν είναι βέβαιη καν αν θα αναλάβει οποιαδήποτε δράση. Δεν είμαι βέβαιος για το τι σκοπεύουν να κάνουν σήμερα. Μα συμφέρει ωστόσο όσοι από εμά πιστεύουμε στην Ευρώπη, είτε είμαστε αεροσκεπτικιστέ ή ε, υπέρ τη Ομοσπονδία, εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην Ευρώπη και η Νορβηγία χρησιμοποιείται ω παράδειγμα για να μην είμαστε στην Ευρώπη. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να μα δώσουν η Κομισιόν κάποια ιδέα, κάποια εικόνα του πώς αισθάνεται, να ρωτήσω ότι να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, τον κύριο Τζον Κλάρκ από την DG Agri. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την ώρα θέλω να πω ότι πρέπει να συγχαρούμε την Νορβηγία διότι έχουν επιτύχει το αδύνατον. Συνένωσαν και κατάφεραν να συμφωνήσουν μεταξύ τους στο Συμβούλιο, η και το Κοινοβούλιο κατά αυτών των περιορισμών. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το σχέδιο ψηφίσματο. Συμφωνούμε με τη θέση τη Επιτροπής και τι απόψει που εκφράζονται σε αυτό το ψήφισμα και τι ανησυχίε για αυτά τα μέτρα. Όπω και εσεί, η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτά τα μέτρα είναι προστατευτικά, ότι αυτό είναι ο σκοπό του και το αποτέλεσμά του, Δεν είναι δράσει που περιμένει κανεί από φίλου και γείτονε. Ε, κατά τη δική μα αξιολόγηση, αυτοί οι εμπορικοί περιορισμοί είναι αντίθετοι με τις διατάξει του ΕΟΧ και με το άρθρο 19 της Συμφωνίας για τη Γεωργία που όπως είπε ο κ. Χέλνερ προβλέπει ε, προοδευτική απελευθέρωση και όχι το αντίθετο. Ακόμη και αν είναι μικρή η επίπτωση αυτών των μέτρων ε, στο συνολικό εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας, παρόλα αυτά τα μέτρα αυτά επικεντρώνονται σε ορισμένους εξαγωγούς και σε ορισμένα κράτη-μέλη και συνεπώς είναι επιζήμια για αυτούς η Νορβηγία δεν μας συμβουλεύτηκε καθόλου για την υλοποίηση αυτών των μέτρων και παραβιάζει σαφώ τι υποχρεώσει τη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε και να το καταλάβουμε ή να το εξηγήσουμε. Ακολούθησαν διαβουλεύσει σε τεχνικό επίπεδο, ξενομοθετικό επίπεδο και ο κύριο Μπαρό ο ίδιο και σε πολιτικό επίπεδο. Το συζήτησε ο κύριος Μπαρόζο με τον Πρωθυπουργό τη Νορβηγία τον περασμένο μήνα, αλλά χωρί κανένα αποτέλεσμα. Η Νορβηγία δεν φαίνεται να προτίθεται να αναθεωρήσει τα μέτρα αυτά. Ενώ θα ήταν πολύ απλό για την Νορβηγία εφόσον είχε την πολιτική βούληση. Για παράδειγμα, η τελωνιακή διαβάθμιση ή το επίπεδο δασμών για τις ορτανσίες θα μπορούσε να αναθεωρηθεί και να επανέλθει ο αρχικός δασμός. Δεν είναι δύσκολο να ληφθούν τέτοια μέτρα. Για να απαντήσω τώρα στο ερώτηση του κ. Στέρντι εμείς τώρα εξετάζουμε τις ε, νομικέ μας επιλογές, ε, τι είδου νομική προσφυγή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν είναι επιλογή, όπως αναφέρει το ψήφισμα, αλλά διμερό. εξακολουθούμε να αξιολογούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εγώ μάλλον συμφωνώ με το αίσθημα αυτό που εκφράζεται στο ψήφισμα, ότι θα έπρεπε να επιλέξουμε αναθεώρηση του πρωτοκόλου και να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει με την Νορβηγία για περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου, μέσω τη οποία θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση για αυτό το πρόβλημα. Προτιμώ αυτή την προσέγγιση, αντί για αντίπεινα ε, εμπορικά, με περιορισμού των εμπορίου. Αλλά πρέπει να πω ότι αν δεν αρθούν οι περιορισμοί αυτοί, την ημέρα που θα στραφεί προς εμάς η Νορβηγία και θα μας ζητήσει την καλή μας βούληση και τη βοήθειά μας, θα το λάβουμε αυτό το συμβάν που βλέπουμε τώρα υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω ξανά το... Πριν δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Φιέλνερ, θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ έχω την αίσθηση, κύριε Φιέλνερ, ότι το ζήτημα αυτό είναι σοβαρό. Δεν είναι μόνο κίνηση που δεν θα έπρεπε να προέρχεται από φίλο, δεν θα έπρεπε να προέρχεται και από γείτονα, από μια γειτονική φιλική χώρα. Και ε, δεν μπορούμε να καταπολεμάμε μέτρα προστατευτισμού στην Αργεντινή και στη Ρωσία και να επιτρέπουμε ταυτόχρονα σε μια γείτονα χώρα, φίλη, να υιοθετεί τέτοια μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα ισχυρό και ενωμένο μήνυμα στο Όσλο είτε να αναθεωρήσει αυτά τα μέτρα ή διαφορετικά θα χρειαστεί να διατρέψουμε σκληρή τάση με την Νορβηγία. Κύριε Φιέλνερ, ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποτέ δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα κανένα προστατευτή, κανέναν να το λέω αυτό, αλλά πολύ κόσμο που αισθάνεται την ανάγκη να πάρει προστατευτικά μέτρα για προστατευτική. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται τώρα. Έχουμε με τους ε, ε, Νορβηγοί Πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με το συναδέλφους του Κοινοβουλίου της Νορβηγίας. Ε, δεν έγινε η πρόταση για αυτά τα μέτρα από τους πολιτικούς ε, και τους κοινοβουλευτικούς στην Νορβηγία και βεβαίως εδώ πλήττονται οι καταναλωτές. Χαίρομαι που είπε η Επιτροπή ότι κατόρθασε η Νορβηγία να δημιουργήσει κάποια πολιτική συνένεση, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει σε σχέση με το θέμα αυτό πολιτική συνένεση Νορβηγία. Γίνονται μεγάλες συζητήσεις και όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι σημαντικό να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Και πρόκειται για ένα πολιτικό μήνυμα, το οποίο βεβαίως στέλνουν οι πολιτικοί με τον τρόπο ενεργών. Τελειώνοντας θα πω... Έχουμε ακόμη την δυνατότητα να κάνουμε κάτι το θετικό. Δεν είναι το τέλος της όλης ιστορίας. και ελπίζουμε ότι ίσως αυτό το πράγμα που με την Νορβηγία έρθει ως κάτι το αρνητικό μπορεί να γίνει κάτι το πιο θετικό. Να συζητήσουμε για τις εμπορικέ ε, ε, σχέσεις μας γενικότερα και όπως είπε η Κομισιό, να αρχίσουμε βάσει της υπάρχουσας συμφωνίας που υπάρχει στα πλαίσια του ΟΧ κάποιες συζητήσεις για τις εμπορικές μας σχέσεις Και θα πρέπει στα πλαίσια της απελευθέρωσης να δούμε πόσο μας ενδιαφέρει ένθεν και ένθεν να ανοιχτούμε περισσότερο. Εάν μπορούσαμε λοιπόν αυτή την αρνητική περίπτωση να την κάνουμε κάτι το θετικό, θα υποφεληθούμε και η μεν και η δε. Και τελικά, συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ίσως θα μπορούσαμε κάτι το αρνητικό να το κάνουμε κάτι το θετικό. Και αν εμεί συνεισφέρουμε για να γίνει θετική όλη αυτή η ιστορία, πάλι καλά. Μακάρι, μακάρι όπω λέτε κι εσεί. Ελπίζουμε ότι όμως και θετικά μηνύματα θα φτάσουν για το Όσλο. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. τη 25 Μαρτίου, σε 5 μέρες, στις 6 το απόγευμα. Και η προφορική αυτή ερώτηση θα συζητηθεί και από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Περνούμε τώρα σημείο 10. Η πρόοδος των τριμερών διαπραγματεύσεων. It is an not a group. Συγγνώμη, συγγνώμη. Επί της ουσίας η ίντα είναι υπεύθυνη. Με συγχωρείτε, λέει πρόεδρος, εγώ έκανα λάθος προηγουμένως. Δεν το... Δεν είναι θέμα πολιτικών ομάδων. Λοιπόν, Σημείο 10. πρόοδο των τριμερών διαπραγματεύσεων. We have uh, not less than four ongoing trilogues. Τέτοιου είδους τριμερείς διαπραγματεύσεις, ε, ε, διαπραγματεύσεις τη στιγμή γίνονται σε τέσσερα. Δηλαδή, είμαστε νομοθετικά μια πάρα πολύ δυναμική και ενεργός επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο θέμα αφορά τις μακροχρηματοπιστωτικές τον κανονισμό πλαίσιο για τις μακροχρηματοπιστωτικές ενισχύσεις. Στις 27 Φεβρουαρίου έγινε πρώτη συνάντηση. Ο κύριος Μετ είναι ο δικός μας εισηγητής ο οποίος σήμερα δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά εγώ ήμουν παρόν και ηγήθηκα όλων των συνεδριάσεων που έγιναν σε τριμερές επίπεδο και παρακολούθησα τις συζητήσεις. Uh, Θα μπορούσα να σας αναφέρω την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και ποια είναι τα κυριότερα θέματα τα οποία παραμένουν εκκρεμή και πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω με το Συμβούλιο. Στην τελευταία τριμερή συνάντηση σημειώθηκε πρόοδος σε διάφορα αμφιλεγόμενα και εκκρεμή θέματα και είμαστε στα πρόθυρα της συμβαστική Τα κύρια θέματα τα οποία ακόμη παραμένουν προς συζήτηση αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία υιοθέτηση του μνημονίου μεταξύ όλων των ε, δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τα θέματα επιτροπολογίας. Στην ε, επόμενη συνάντηση θα συζητήσουμε και το θέμα των κατοφλίων. στα οποία θα κινηθεί το μνημόνιο. Πρέπει να πω ότι υπάρχει σημαντική σύγκληση απόψεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αλλά δεν συμφωνεί η Επιτροπή. Δεν συμβαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη φορά έχουμε από τη μια μεριά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και από την άλλη την Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκφράζουν τη λύπη τους διότι η απόφαση για την χορήγηση βοήθεια σε τρίτες χώρες θα εγκριθεί σύμφωνα με την συνήθη διαδικασία, τη συναπόφαση δηλαδή, μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής, ενώ η Επιτροπή εμένει στην αρχική της πρόταση ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται βάσει πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Το δεύτερο σημαντικό θέμα, όπως ήδη σας είπα, η επιτροπολογία. Και εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ αφενός του Κοινοβουλίου και αφετέρου του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο επιμένει στην διαδικασία βάση της οποίας έχουν το δικαίωμα άρνηση κυρίας Βέτο τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, δυνατότητα εφαρμογής των αποφάσεων Εγμένης Επιτροπής. Μιλώ πάντα για την ε, χρηματοπιστωτική ενίσχυση. Λέμε ότι θα πρέπει να εγκριθεί βάση της συνήθως διαδικασίας. Ίσως ο συμβιβασμός θα είναι να έχουμε και πάλι ένα κατόφλι για την ενίσχυση και ανώτερα ποσά θα εξεταστούν, θα προταθούν και θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Και θα επιτραπούν κάποιες εξαιρέσεις. για κάποιες αποφάσεις που αφορούν την ε, χρηματοπιστωτική ενίσχυση. Αν φτάσουμε σε συμφωνία θα τηρήσουμε τους ισχύοντες κανονισμούς. Θα δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες βάσει της νομοθεσίας, πώς θα χορηγηθεί η ενίσχυση στις τρίτες χώρες. Και η απόφαση θα ληφθεί βάσει της ε, ε, νομοθεσίες της συνήθως, δηλαδή θα έχουμε την νομοθεσία πλαίσιο και μετά τους διάφορους κανονισμούς βάσει των οποίων θα χορηγηθεί αυτή η χρηματοπιστωτική ενίσχυση. Uh, the, state of the uh, play. Let's see what the next... Αυτό είναι το έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει στα πλαίσια τη επόμενη συνάντηση, τριμερού διαλόγου. ίσως καταλήξουμε και σε συμβασμό μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Τώρα, για το Omnibus 1. Στις 5 Μαρτίου έλαβε χώρα ο τελευταίος τριμερής διάλογος. Εισηγητής. Ή η συγγετρή κυρία Κίσταουτ δεν είναι εδώ. Αλλά αφού ήμουν εγώ εκεί, μπορώ να σας ενημερώσω για το τι ακριβώς έγινε. Τα θέματα σε κρεμότητα είναι λίγα. Υπάρχει σύγκληση απόψε μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την πρόταση επιτροπής. Έκρεμη θέματα είναι η διάρκεια της νομοθετικής εξουσιοδότησης που θα δοθεί στην Επιτροπή, η χρονική προθεσμία για να υπάρξουν αντιρρήσεις, τρίτον το Κοινοβούλιο δικαιούται να συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων για την προετοιμασία των πράξεων κατά εξουσιοδότηση και κάποια θέματα που αφορούν την επιτροπολογία. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις από το Συμβούλιο ότι μπορούμε ίσως να επιτύχουμε για τα θέματα ακόμη που δεν έχουν επιληθεί συμβιβαστικές λύσεις, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε δεδομένο. Θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη συνάντηση σε τριμερές επίπεδο για να δούμε αν πραγματικά θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένε συμβαστικέ λύσει. Έχω παρόλα αυτά την εντύπωση ότι η Ιρλανδική Προεδρία στον τομέα αυτό έχει να παρουσιάσει νέες ιδέες, τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω. Είναι ντροπή το ότι φτάνουμε στο τέλος της παρούσης θητείας χωρίς να έχουν γίνει οι προσαρμογές του νομοθετικού κεκτημένου. Τώρα, Omnibus 2, που είναι ο άλλος κανονισμός που αφορά τον νομοθετικό κεκτημένο τη ε, κανονισμούς επιτροπολογίας. Ο κύριος Λάιφριντ είναι εισηγητή. Δεν είναι παρόν, εγώ όμω ήμουν και άρα μπορώ να σας ενημερώσω και τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο. Και αυτή τη φορά έχω κάποιο σημείο που μου στείλει ο εισηγητής για το θέμα αυτό πρώτη συνάντηση τριμερής επίσης έλαβε χώρα στις 5 Μαρτίου και οι σκιώδεις ε, οι συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. τεχνική συνάντηση θα λάβει χώρα αυτή την Παρασκευή και δεύτερη συνάντηση σε τριμερές επίπεδο θα γίνει τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Πρόκειται για παράλληλο φάκελο με αυτό του Omnibus 1 και τα εκκρεμή θέματα είναι τα ίδια με το Omnibus 1. Και συμφωνήσαμε ότι παρά το γεγονός ότι γίνονται διαφορετικές συνεδριάσεις, θα πρέπει να γίνονται με συντονισμένο τρόπο και εκ παραλίλου. Είμαι σίγουρος ότι με τους ε, δύο συντονιστές θα επιτευχθεί ο συντονισμός και στο τέλος θα καταλήξουμε σε συνεκτικά αποτελέσματα. Όπως ήδη σας ενημέρωσα και για το Omnibus 1, έχω την εντύπωση ότι η Ιρλανδική Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία και για αυτό το θέμα. Καλό θα είναι, καλό θα είναι αυτό για την Προεδρία αυτή. Ε, έχετε κάνει μια ερώτηση. Ξέχασα να σας ρωτήσω αν έχετε μετά από όλα αυτά τα οποία είπα ερωτήσεις να κάνετε. Δεν βλέπω κανένας να θέλει να κάνει ερωτήσεις. Και τελικά... τέταρτος και πιο σημαντικός ε, φάκελος, πρόσβαση στην αγορά. Προθεσμία για την υπογραφή και επικύρωση ε, της, ε, των εμπορικών ε, συμφωνιών με τις χώρες ΑΚΕΜ. Όπως ξέρετε, σύμφωνα με τη Συμφωνία της Κοτονού υπάρχουν κάποιες προτιμήσεις, προτιμησιακές συμφωνίες, οι οποίες δεν συμφωνούν με τους αποφάσεις επίπεδο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα πρέπει να υπογραφούν και να επικυρωθούν συνολίες, ώστε να μην ε, χάσουν αυτή την προτιμησιακή ε, μεταχείριση οι χώρες αυτές. Στις 6 ε, Μαρτίου είχαμε δεύτερη συνάντηση. Ο David Μάρτιν, ο εισηγητής, είναι παρόν. Εθημέρωσέ μας λοιπόν εσύ για τις τελευταίες εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε τα βασικά, οπότε θα είμαι σύντομος. Υπήρχαν τρία διαφορετικά ζητήματα που έπρεπε να δούμε. Το πρώτο ήταν εύκολο και ξεκαθάρισε γρήγορα. Ήταν καθαρά γλωσσικές αλλαγές που ήθελε να κάνει το Συμβούλιο που δεν επηρέαζαν την ουσία, οπότε ευχαριστώ τις δέχτηκα. Το δεύτερο αφορούσε διατάξεις τύπου επιτροπολογίας όπου είχαμε τρεις ε, τροπολογίες ε, στην έκθεση. Το Συμβούλιο ήταν διατεθειμένο να δεχτεί μία από τις τροπολογίες ε, που αφορούσε χώρις εξουσιών για πέντε έτη με δυνατότητα ανανέωσης μόνο αν το δεχόταν το Συμβούλιο. Για τις άλλες δύο διατάξεις επιτροπολογίας συμφωνήσαμε να μην αλλάξουμε την θέση μας, αλλά να μην επιμείνουμε γιατί είχαν αντιμετωπιστεί αυτά τα ζητήματα στο Omnibus 2 και είχαμε κάνει αρκετά καλή πρόοδο. Το βασικό ζήτημα βεβαίως ήταν η ημερομηνία που εμείς στο Κοινοβούλιο θέλαμε την 1η Ιανουαρίου 2016 το Συμβούλιο υποστήριζε την θέση της Κομισιόν για το 2014. Ήταν δύσκολες διαπραγματεύσεις γιατί η Προεδρία είπε πως είχαν εντολή να πάνε μόνο μέχρι την 1η Ιουνίου 2014 που ήταν απαράδεκτο για εμάς. Η δική μου η άποψη και ίσως προδόθηκα ήταν πως θα έχουμε κάποιον συμβιβασμό ε, και ανέμενα την 1η του 2015. Τελικά αυτό δεν έγινε και πήγε πέρα από τον Ιόνιο το Συμβούλιο και Φτάσαμε στην 1η Οκτωβρίου 2014. Δεν είναι ιδεώδης η ημερομηνία, αλλά είναι ό,τι καλύτερο θα επιτύχουμε. Οπότε δέχτηκα το αποτέλεσμα του τριμερού διαλόγου και την 1η Οκτωβρίου 2014 ως την ημερομηνία στην οποία θα τελειώσει η πρόσβαση στην αγορά. Μάλιστα. Είχαμε έναν συμβιβασμό λοιπόν και θα ψηφιστεί αύριο. δεύτερη ανάγνωση είναι, οπότε χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Οπότε στα από τις πολιτικές να είναι παρούσες αύριο για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ήμουν μέλος της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας και είχα εμπλακεί στο ζήτημα του πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο επικοδομητική διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θέλω να παρατηρήσω πως ε, δεν βρήκα πάρα πολύ ευνοϊκό το ότι η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία δεν προσπάθησε μέχρι το τέλος να περάσει ως κοινή γραμμή την γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δόθηκε ως μήνυμα στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο, όπως η απόφαση της Ολομέλειας του Στρασβούργου ε, μπορούσε και να μην ε, υποστηριχθεί εντελώ. Και άρα εξασθένησε η διαπραγματευτική μας θέση. Αύριο λοιπόν που θα ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες, τις ημερομηνίε και ο Ντέιβιντ Μάρτιν τα είπε ξεκάθαρα, πρέπει να σκεφτούμε μήπως έχοντας κατά νου τις πολιτικές διαδικασίες της χώρας εταίρους εδώ πέρα, μήπως να προσπαθήσουμε να έχουμε μια διαφορετική τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέσο αυτό. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ας θυμηθούμε τα βασικά. Όταν ε, έχουμε μια διαπραγματευτική θέση στην Ολομέλεια, ε, είναι μια εντολή για διαπραγμάτευση, αλλά εξυπονοείται πως υπάρχει κάποια ευελιξία, έτσι αλλιώς δεν υπάρχει λόγος ε, διαπραγμάτευσης. Θα έλεγε ο καθένας ε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο στον άλλον τη θέση του και βεβαίως όλες οι συμβαστικές προτάσεις είναι αντρεφερέντουμ, δηλαδή πρέπει να επανέλθουν στην Επιτροπή για να κυρωθούν. Αυτό το οποίο κάναμε λοιπόν ε, είναι ακριβώς αυτό το οποίο είχαμε κάνει σε οποιοδήποτε ε, τριμερή διάλογο. Δηλαδή εγώ, οι συγητές και οι σκιώδες συγητές θεωρούν πως έχουμε μια εντολή να παλέψουμε, αλλά στη διαπραγμάτευση μπορούμε να έχουμε κάποια ευελιξία για να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό. Ό,τι άποψη και να έχουμε, και, και εγώ βεβαίω έχω κάποια προσωπικά συναισθήματα, γιατί ήμουν εκεί συμμετείχα στο ημερή διάλογο. Θεωρώ πως ήταν η καλύτερη συμβαστική λύση που μπορούσαμε να επιτύχουμε. Είχαμε κερδίσει τους 9 μήνες, όχι τα, τα τρία χρόνια που θέλαμε. Τέλος πάντων, κάτι έγινε και Θεωρούσαμε πως το Συμβούλιο δεν είχε περιθώριο να προχωρήσει παραπέρα. Και η 1η Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία γιατί τότε λίγη η θητεία της Επιτροπής μας και ε, ήταν σαφές πως δεν θα μπορούσε η Κομισιόν να επιτρέψει το φάκελο αυτό να περάσει στην επόμενη Επιτροπή. Οπότε αύριο η Επιτροπή μας θα πρέπει να κυρώσει τα όσα είναι. Όπως είπα, όλοι οι συμβασμοί είναι ad referendum. είναι μια φράση στα λατινικά που σημαίνει θα παραπεμφθεί σε κάποιον. Έτσι. Και θα κρυφθεί από αυτόν. Οπότε ε, δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση εδώ πέρα κάτι διαφορετικό. Οι φιλελεύθεροι θέλουν να πούν κάτι. Ναι. Εγώ έχω τις ίδιες απόψεις με εσάς και τους συναδέλφους της Επιτροπής όπως είπατε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις μερικές φορές δεν κερδίζουμε όσα θα θέλαμε και αυτό είναι κρίμα, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την αιμονή του και την εξαιρετική του δουλειά. Πιστεύω ωστόσο ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε με την ψηφοφόρη αύριο και με βέβαια ότι μπορούμε να δεχτούμε ε, τις συστάσεις του εισηγητή, αλλά πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα από όλα αυτά. Έχουμε παρακολουθήσει και βέβαια στο μεταξύ έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουμε, αλλά εδώ και χρόνια παρακολουθούμε διαπραγματεύσεις άσκοπες που δεν πηγαίνουν προς τα πουθενά και ξαφνικά πέφτει η προθεσμία του ενός έτου. Ε, όπου πρέπει να ολοκληρώσουμε και δεν μου φαίνεται ότι αυτός είναι φυσιολογικό τρόπο διαπραγματεύση με ισότιμους εταίρους ε, πνεύμα δικαιοσύνη και καλή διάθεση. Πιστεύω ότι Ελπίζω μάλλον ότι η Κομισιόν έχει λάβει τα μαθήματα του πώς πρέπει να διαπραγματεύεται, ειδικότερα με αναπτυσσόμενες χώρες που δεν νιώθουν ισότιμοι εταίροι στις διαπραγματευτικές ομάδες. Έχουμε προθεσμίες, ε, ξέρουν ας πούμε ότι έχουμε δύο χρόνια για να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις, διότι Αλλιώ βρισκόμαστε σε μια δυστυχή κατάσταση. Εργότερα αυτή τη εβδομάδα έχουμε τη συνάντηση τη Επιτροπή ACP και πολλά μέλη από αυτέ τι χώρε θα βρίσκονται εδώ και θα παρακολουθούν τι θα κάνουμε και αύριο και θα πρέπει αργότερα μέσα αυτή την εβδομάδα να του εξηγήσουμε γιατί βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Είναι ένα δυστυχέ επεισόδιο και ελπίζω να μάθαμε το μάθημά μα και ε, όσοι διαπραγματεύονται, είναι διαπραγματεύονται εκ μέρου εμά ε, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν μάθει κάποιο μάθημα, κάποια ε, δεξιότητες διαπραγμάτευσης ε, καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος. Να απαντήσω σε αυτό το οποίο είπε η συνάδελφος. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση γιατί μιλάμε με κάποιες χώρες για ένα θέμα το οποίο προφανώς ε, αντιβαίνει τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτό ε, δεν έγινε χτες ή σήμερα αντίθετο με τους κανόνες του ΠΟΕ, αλλά προ, προ, προ, χτες. Και είχαμε 10 χρόνια στη διάθεσή μας να κάνουμε κάτι. Τώρα είναι ε, περίεργο να κατηγορούμε και την Κομισιόν για το ότι δεν υπήρχε ε, αποτέλεσμα. Γιατί έρχονται και σε μένα κάποιοι και μου λένε το κοινοβούλιο φταίει. Γιατί υπάρχουν πάντα κάποιοι ευρωβουλευτές οι οποίοι ε, λένε πως ε, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο και ας τα αφήσουμε κάνα δύο χρόνια ακόμα για τις διαπραγματεύσεις και, έτσι δεν καταλήγουμε πουθενά. Και αν δεν γίνει τίποτα θα φροντίσουμε να παραμείνει η κατάσταση όσο έχει μέσω του Κοινοβουλίου. Τώρα δεν ξέρω λοιπόν αν η Κομισιόν έκανε λάθος διαπραγματευσία αν έστειλε λάθος μήνυμα το Κοινοβούλιο. Πρέπει να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Η ίδια ομάδα μου θεωρεί πως πρέπει να περάσει αυτός ο συμβασμός από το Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να πω πως αν δεν έχουμε κάποια πλειοψηφία, τότε ε, θα επιμείνουμε σε αυτά τα οποία είχαμε πει ε, στην Ολομέλεια. Είναι, είναι μια απλή διαπίστωση. Έτσι. Γιατί θεωρούμε πως είναι καλός ο συμβασμός. Τώρα αν είναι 1η Ιανουαρίου 2015 ή 1η Οκτωβρίου 2014, ε, τώρα για αυτούς τους λίγους μήνες δεν πρέπει να το καταστρέψουμε αυτόν τον συμβασμό. Όλοι δεν μας είπαν στις χώρες μας πώς επιθυμούν να ολοκληρωθούμε να ολοκληρωθεί κάποτε αυτή η διαδικασία που κρατάει σχεδόν 10 χρόνια. Πρέπει επιτέλου να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Είναι και αντίστοιχο με του κανόνε του ΠΟΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ντάνιελ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον Ντέιβιντ. Διότι πιστεύω ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα και στις δύο περιπτώσεις. Ήταν σχεδόν μια δύνατη κατάσταση. Άλλοι ήθελαν μια ημερομηνία αργότερα, άλλοι νωρίτερα. Είναι ένα συμβιβασμό και οι συμβιβασμοί Ποτέ. Δεν ικανοποιούν όλους. Διαφωνώ όταν λέτε ότι τους το πετάξαμε. Έτσι ξαφνικά το γνώριζαν εδώ και καιρό ότι αυτό θα αποφασιζόταν αργά ή γρήγορα. Η απόφαση ελήφθη. Εγώ συμφωνώ με την απόφαση αυτή γιατί πιστεύω ότι καθαρίζει, ξεκαθαρίζει τα πράγματα και τους επιτρέπει να προχωρήσουν και να κάνουν ό,τι χρειάζεται να κάνουν. Εγώ νομίζω ότι πράξαμε σωστά και ο συμβιβασμός είναι αποδεκτός για τη δική μου ομάδα και πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη τελική συμβαστική απόφαση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος Φρανσίσκη Γκέλλερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να πάψουμε να συζητάμε το περιεχόμενο. Έχουμε προσθέσει όλα τα επιχειρήματα. Έχουμε ανταλλάξει όλα τα επιχειρήματα πριν την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Άλλοι ήθελαν να υπάρχει συντομότερη επιθεσμία, άλλη μεγαλύτερη και εν τέλει στην Επιτροπή ψηφίστηκε μια τροπολογία με την πλειοψηφία αυτή τη Επιτροπή. Συνεπώ αυτό αποτελεί απόφαση του Κοινοβουλίου. Θέση του Κοινοβουλίου και αυτή η θέση του Κοινοβουλίου ε, σύμφωνη με τη θέση του Συμβουλίου επειδή είμαστε συνομοθέτες και μάλλον δεν συμφωνεί απόλυτα με το Συμβούλιο. Οπότε μπορεί να καταλήξουμε σε μια συμβιβασμό και των δύο αυτών πλευρών. Πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση το Κοινοβούλιο σαφώ υποχώρησε. Πιστεύω ότι είναι κακή, κακό συμβιβασμό. Διότι απόψη διαδικασία θα πρέπει να προσπαθούμε να υπερασπιζόμαστε τη θέση του Κοινοβουλίου, ακόμη και αν είναι η δική μα προσωπική θέση, για να διατηρήσουμε και την αξιοπιστία αυτού του Κοινοβουλίου. Εγώ συμμετέχω σε πολλέ τριμερεί διαπραγματεύσει όπου έχω Ήδη χάσει πολλά, αλλά παρόλα αυτά, ε, ή δεν συμφωνώ με τη θέση της ε, Επιτροπής, αλλά εγώ στηρίζω την τη θέση του Κοινοβουλίου, γιατί αυτή είναι η θέση μας ως συνομοθέτης. Αν χάσουμε την αξιοπιστία μας, αν δεν είμαστε ενωμένοι και δεν στηρίζουμε ενωμένοι τη θέση του Κοινοβουλίου, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καλά, γιατί θα έχουμε προβλήματα και σε άλλες τριμερείς διαπραγματεύσεις με διαφορετικές πλειοψηφίες εντός της Επιτροπής. Τώρα, για να σας απαντήσω, λέει ο Πρόεδρος, δεν πιστεύω ότι υπάρχει απώλεια αξιοπιστία του Κοινοβουλίου. Εδώ ψηφίστηκαν δύο ζητήματα. Και με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε αυτό. Και μάλιστα οι πράσινοι ψήφισαν κατά. Αυτή ήταν η απόφαση κλειδί. Το κατά πόσο πρέπει να υπάρχει προθεσμία. Και η προθεσμία ήταν είτε το 2013 είτε το 2013. Και ο συμβιβασμό πέφτει στη μέση. Συνεπώς δεν έχει υποχωρήσει το Κοινοβούλιο. Κέρδισε ένα συμβιβασμό. Μην ε, λέμε λοιπόν τέτοια πράγματα. Δεν υπήρξε υποχώρηση και καμία απώλεια αξιοπιστίας. Κάναμε ό,τι κάνουμε πάντα. Κάθε φορά. Έχουμε μία εντολή, αλλά ευέλικτη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού. Αυτό παρουσίασε και ο εισηγητή και εγώ σε αυτή την επιτροπή. Είτε επικυρώνουν οι άλλοι, είτε λένε όχι. Οι πράσινοι μπορούν να ψηφίσουν κατά, έχουν την ελευθερία να το πράξουν. Αλλά όχι λόγω της προθεσμίας. είστε κατά οποιασδήποτε προθεσμίες, όχι αυτή τη προθεσμία γιατί ψηφίσατε κατά. είμαστε λοιπόν ειλικρινεί. Είναι δύο πολύ διαφορετικά ζητήματα. Το δεύτερο είναι δευτερεύον το ζήτημα κλειδί αποφασίστηκε από μεγάλη πλειοψηφία σε αυτή την Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Και οι πράσινοι ψήφισαν κατά. cannot allow Δεν μπορώ να επιτρέψω να αμφιβάλλουμε ανετιολόγητα την αξιοπιστία αυτού του κοινοβουλίου. Να την αμφισβητούμε. Ήμουν παρόν. Σημείο 11. Δραστηριότητες εποπτικών ομάδων. Από τις... Υπάρχουν πολλές εποπτικές ομάδες η ομάδα για τη Ρωσία είχε μια συνεδρία πρόσφατα στις 7 Μαρτίου και δίνω το λόγο στον συγκεκριτή, στον Ρομπερ Σέρντι. Δεν μπόρεσα να είμαι παρόν, ο Τζόρτζ ήταν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια μόνο. Ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες παρακολούθησης που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ποιο λόγο? διότι στην ομάδα παρακολούθησης είχαμε τον κύριο Τίμασμαν, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι νομικός, έχει μεγάλη εμπειρία με τη Ρωσία, επειδή αντιπροσώπευσε τους ε, επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου στη Γιούκος και εγώ θα του συνέστηνα να γράψει ένα βιβλίο για τις εμπειρίες του με τη Ρωσία. αποτέλεσε πολύ καλό διάδραμα για την Κομισιόν, μάθημα για την Κομισιόν, ας πούμε, διότι είναι απίστευτο. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ίσως υπό άλλες περιστάσεις θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Αλλά, όπως είπα, ήταν πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι για το μέλλον της μελλοντικέ διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία είναι σημαντικό να μάθουμε από τις εμπειρίες ε, του παρελθόντος και ελπίζω, Ρόμπερτ, ε, επειδή είσαι εισηγητής, ε, πιστεύω ότι αυτού του είδους οι εμπειρίες ε, καλό είναι να επαναληφθούν πολλάκις. Σίγουρα η Ρωσία είναι ενδιαφέρον για εμάς, θέλουμε να είναι εταίρος μας. Δυστυχώς όμως το παιχνίδι που παίζουν είναι ένα εγωιστικό παιχνίδι και δεν ξέρω με ποια λύση θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Είμαι αισιόδοξο εγώ, αλλά δυστυχώς ε, οι ενδείξεις, ε, τα μηνύματα από τη Ρωσία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ευχαριστώ. Σχόλια. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα δεν ήμουν παρόν. Η επόμενη ομάδα παρακολούθησης αφορά την ε, Γεωργία και κάποια άλλα ζητήματα. Ε, όχι την Κύπρο, περιέργως. Ε, αυτά ε, είναι τα σχόλια που έχω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχα την ευκαιρία και εγώ να είμαι παρόν κάποια στιγμή καλύψαμε και το ζήτημα της ενεργειακής συνεργασίας και η τιμή της ενέργειας και αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι πως υπήρχε η άποψη που χράστηκε και από την Κομισιόν πως με ένα κάπως ε, έτσι διαφορετικό τόνο πως ε, η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένα ουδέν σχόλιον. Οπότε πρέπει να δούμε το τι θα κάνουν οι τις διαφορετικές ε, θέσεις των κρατών μελών απέναντι στη Ρωσία και την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να δούμε και το μήνυμα που θα στείλουμε στην ομάδα αυτή παρακολούθησης για να ζητήσουμε τα αποτελέσματα της ε, πρόσφατης συνόδου όπου είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αλλά νομίζω πως πρέπει να συζητήσουμε τις εμπορικές πτυχές για στο πλαίσιο μιας γενικότερης επανεξέτασης της ε, λεγόμενης στρατηγικής σχέσης με την ε, Ρωσία. Εγώ είμαι υπέρ, αλλά αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχουμε και μια κοινή θέση. Οπότε μπορεί να υπάρξει και μια συζήτηση για την πι... ε, για το πώς ε, μεταφέρουμε τις θέσεις μας στη διαπραγμάτευση σε διαφορετικά επίπεδα για να μπορέσουμε πραγματικά να συνεισφέρουμε στη στρατηγική εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, λάβουμε υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στα ενεργειακά, γιατί ειδικά το τι έγινε στην δεύτερη θητεία Ομπάμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, σκοπεύουν να επιτύχουν μια ενεργειακή ανεξαρτησία. Οπότε θα βγάλουν πετρέλαιο και αέριο από την ε, Αλάσκα, από την Αλμπέρτα, στον Καναδά ε, νέοι πόροι στον κόλπο του Μεξικού και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να επιτύχουν μια ενεργειακή ανεξαρτησία και αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγές ενεργειακές αγορές, ειδικά οι χώρες του κόλπου στην ε, Μέση Ανατολή θα στραφούν προς την Ευρώπη ως ε, μια πάρα πολύ καλή αγορά και προς την Κίνα και θα υπάρχει άρα ανταγωνισμός μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και των χωρών της Μέσης Ανατολής ε, στο θέμα αυτό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη μεταβολή για την ενεργειακή πολιτική μας και πρέπει να πω πως εάν συγκρίνουμε την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ομολογήσουμε πως οι ΙΠΑ έχουν μια πραγματική ενεργειακή πολιτική. Δεν σημαίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δικός μας χάρτης για το 2050 είναι μόνο το άθροισμα ευσεβών πόθων και κάποιων ιδεολογιών. Όχι εφικτές και πραγματικές ε, των ενεργειακών μας προβλημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Να τονίσω κάτι το οποίο ακούστηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, από τον συνάδελφο. Δεν πρέπει να έχουμε μόνο κοινή θέση, αλλά να την εκφράσουμε. Ε, εγώ ήμουν επικεφαλής αντιπροσωπείας αυτής της Επιτροπής στη Ρωσία αρχές Οκτωβρίου πέρσι και είχαμε ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου που ευθύθηκε στην Επιτροπή μας και βεβαίως θέλαμε πάρα πολύ να ε, επιμείνουμε σε αυτά τα οποία έλεγε το ψήφισμα και ήταν κάπως περίεργο να ακούμε από τους συναδέλφους μας να μας λένε «Μα αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου, εμείς ξέρουμε πως δεν είναι η θέση όλων των θεσμικών οργάνων είναι ατυχές». Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα με τη Ρωσία. Οπότε νομίζω πως ε, είτε μιλάμε για ενέργεια, την Gazprom, ε, την ιδιοκτησιακή αποδέσμευση, ζητήματα αντιτράστ, ε, ανταγωνισμού που αφορούν την Gazprom ή άλλα ζητήματα. Η μη σεβασμού των δεσμεύσεων απέναντι στον ΠΟΕ. Νομίζω πως πρέπει να έχουμε μια κοινή θέση σκληρή κατά την άποψή μου απέναντι στη Ρωσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημείο 12. Το επόμενο σημείο, το 12. Διαπραγματεύσει σχετικά Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση είπα για το εμπόριο και τι επενδύσει. Είμαστε επί τη ουσία υπεύθυνη Επιτροπή, εγώ είμαι ο εισηγητής, όπως γνωρίζετε η Επιτροπή συμφώνησε στις 12 Μαρτίου να εγκρίνει την ε, εντολή, το σχέδιο εντολή σχετικά με τις προσεχείς διαπραγματεύσεις να αρχίσουν σε επίδοση συμβουλή οι διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή μας αποφάσισε να κάνει ένα ξεχωριστό ψήφισμα για το θέμα αυτό εκτός από το να εκθέσει που είχαμε εγκρίνει πέρσι τον Οκτώβριο το σχέδιο ψηφίσματος. Το έχετε στους φακέλους σας και ως εισηγητής θα ήθελα να κάνω κάποια επεξηγηματικά σχόλια. Πρώτα απ' όλα, το TTP, TTPAU θα μπορούσε να είναι μια ε, διαφορετική συμφωνία από τις άλλες. Η πιο φιλόδοξη, αν θέλετε. Και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την ε, συμφωνία αυτή ήταν ε, διαφορετικές από τις προηγούμενες. Πρώτα απ' όλα, και από τις δύο πλευρές αποφασίστηκε πριν από ένα χρόνο να συσταθεί μία ψηλού επίπεδου ομάδα εργασίας Σε υψηλό επίπεδο η ομάδα εργασία εργάστηκε για 14 ε, μήνες για να δει κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει μία ευρύτατη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκ με όλες τις διαδικασίες που ακολούθησε και τις συνεδριάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου και από την και πέρσι τον Ιούνιο εγκρίθηκε μία, εγκρίθηκαν διάφορες πρώτες εκθέσεις και τελική έκθεση στους τελευταίους μήνες. Εμείς στην Επιτροπή μας αποφασίσαμε επίσης να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στην όλη διαδικασία και αποφασίσαμε να εγκρίνουμε όπως ήδη σας ανέφερα και μια έκθεση πέρσι τον Οκτώβριο. Βασιστήκαμε στην ε, προσωρινή έκθεση της ομάδας εργασίας του και ζητήσαμε τη συνεργασία άλλων επιτροπών που θα ενδιαφέρονταν ενδεχομένως από για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η έκθεση πρωτοβουλίας εγκρίθηκε στην Ολομέλεια με συντριπτική πλειοψηφία και περιλαμβάνει την ε, άποψη του Κοινοβουλίου, τη θέση, τη τοποθέτηση του για το τι μπορούμε να επιτύχουμε με αυτές τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις με πρωτοβουλία της Επιτροπής, τη έκθεση στην Συμβούλιο για να αποφασίσει. Δεν συμμετέχουμε στις αποφάσεις και σύμφωνα όμως με τη προσωρινή συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, έχουμε πρόσβαση στο ε, σχέδιο εντολής και το Συμβούλιο αποστέλνει τα σχετικά έγγραφα σε μένα και τους συντονιστές. Πρόκειται για εμπιστευτικά ε, έγγραφα περιορισμένης ε, ε, δημοσιότητας πριν να αποφασίσει την εντολή τη διαπραγματευτική, το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν και εμείς έχουμε κάτι. Έχουμε το σχέδιο ψηφίσματο λοιπόν. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν ότι ήδη τον Οκτώβριο έχουμε κρίνει μία λεπτομερέστατη έκθεση και δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα πάντα μια δεύτερη φορά, αφενό και αφετέρου, δεδομένου ότι πρόκειται ε, στις ε, διαπραγματεύσεις έχουμε να κάνουμε με εμπιστευτικά έγγραφα τα οποία δεν μπορούμε, να, τα οποία δεν άμεσα να ε, σχολιάσουμε προς το παρόν, δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε ε, όμως την εντύπωση ότι θα είναι ένα δεύτερο ψήφισμα χρήσιμο για να πούμε τι ακριβώς μας απασχολεί και τι θέλουμε να υπάρχει σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Το Κοινοβούλιο, λοιπόν, παρακολουθεί το περί πρόκειται. Θα δούμε το σχέδιο ψηφίσματος. Αναφερθήκαμε στο ψήφισμα μας το Οκτωβρίου και είπαμε ότι θα πρέπει χωρίς να μπούμε σε τεχνικές ή άλλου τύπου λεπτομέρειες να, που είναι εκτός των δικών μας αρμοδιοτήτων ε, να έχουμε σε αυτό το στάδιο και εμείς να πούμε τις απόψεις μας. Τελική παρατήρηση. Πρόκειται για 100% για μία συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων. Έτσι το εκλαμβάνουμε, αλλά όπως σας είπα, θα υπάρξουν στις διαπραγματεύσεις και διάφορα κανονιστικά θέματα κανονισμοί που θα εφαρμόζονται εγκαρσίως και γι' αυτό το θέμα είπα ότι θα ζητήσουμε και τη συνεργασία των ενδιαφερομένων επιτροπών. Γι' αυτό και πάλι αποφάσισα να καλέσω των προέδρους άλλων επιτροπών ε, έστειλα την σχετική επιστολή όπως το είχα κάνει και για την προετοιμασία της έκθεσής μας τον Οκτώβριο για να συμμετάσχουν στη σημερινή συζήτηση. Και από όσον βλέπω, τουλάχιστον μία από τις επιτροπές αποφάσισε να παρίσταται σε, αυτές, σε αυτή τη συνεδρία σήμερα. Έχουμε λοιπόν μία μνημεμάδα που σχολείται με αυτό το θέμα των διαπραγματεύσεων για το εμπόριο και τις επενδύσεις με τις πριν να αποφασιστούν οι διαπραγματεύσεις. Άρα είμαστε προετοιμασμένοι κατά κάποιο τρόπο και θα δώσω ε, στις συναδέλφους του λόγο. Η κυρία Κουστίδη πρώτα απ' όλα. Έχει το λόγο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως με χαρά διαπιστώνουμε πρώτον πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΙΠΑ θα ξεκινήσουν και θα προχωρήσει η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, τουλάχιστον τα προπαρασκευαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως ε, όλα τα θετικά δεν χρειάζεται να τα ξαναδούμε εκ νέου για λόγους τυπικούς, οπότε θα είμαι σύντομη θεωρώ σωστό εμείς ως Κοινοβούλιο να συντάξουμε ένα δεύτερο ψήφισμα, ακόμα και αν κάποια πράγματα ε, που έχουν ήδη υποθεί επαναληφθούν. Εάν, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ε, είναι να είμαστε σύντομοι, οφείλω να πω πως είναι πολύ μακροσκελές το ψήφισμα. Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε αυτά τα οποία έχουμε ήδη επαναλάβει και να επικεντρωθούμε στα ουσιαστικά. Τα μισά εκτιμώντας δηλαδή μπορούν να φύγουν. Το οικονομικό και πολιτικό, η οικονομική και πολιτική συγκυρία επίσης δεν ωφελεί τίποτα. Ε, σημασία έχει λοιπόν αυτό το οποίο αναφέρεται στα τελευταία σημεία, η διαπραγματευτική εντολή και ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Και έχετε δίκιο όταν τονίζετε πως είναι μία εμπορική συμφωνία. Εδώ πέρα παίζουμε άρα εμείς τον κύριο ρόλο και θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις για τα σημεία 16 και 18. Θεωρώ πως μέσω της ε, διατλαντικής αυτής ε, συμφωνίας έχουμε κάνει τόσο λεπτομερεί λεπτομερείς ε, συζητήσεις ώστε θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα εδώ πέρα, να κάνουμε μια πρόταση δηλαδή τα σημεία 16 και 18 να συνδυαστούν. Θα ήταν πάρα πολύ καλό εκεί όπου υπάρχουν δυσκολίες με προδιαγραφές κτλ. Οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά δουλεύουν με αυτά τα ζητήματα να είναι μαζί μας στο τραπέζι και είτε να ε, εκπροσωπηθούν στην ομάδα διαπραγματευτική της Κομισιόν του Κοινοβουλίου για να έχουμε και την άποψη ανθρώπων που ασχολούνται με τα ζητήματα πρακτικά. Επίση, για τον ρόλο του Κοινοβουλίου ε, συμφωνούμε ευτυχώ επί τη ουσία και για το σημείο 22 θα πρέπει να συνεργαστούμε εντατικά με Συμβούλιο Κομισιόν, Κογκρέσο κτλ. Και εγώ θα προσέφετα πως πρέπει αυτό να γίνει σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Γνωρίζουμε πως ε, αυτή τη έχουμε μία νομοθεσία ε, που θα πρέπει να περάσει σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να έχουμε κύρωση από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Οπότε, αν είναι να μιλάμε για αποδοχή από την κοινή γνώμη στην κάθε χώρα και στην κάθε πρωτεύουσα, καλό θα είναι και οι εθνικοί συνάδελφοι, ε, βουλευτές δηλαδή, σε τακτά χρονικά διαστήματα να συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία. Μια τελευταία παρατήρηση που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σχέση με το ψήφισμα αυτό, είναι σωστό να το ότι λαμβάνουν οι συντονιστές το κείμενο, αλλά θα ήταν απλούστερο να έχουν και τα κείμενα των συντονιστών. Είναι νομίζω κάτι το απλούστερο από το να ε, κάνουμε όλες αυτές τις διαδρομές. Βεβαίως αντιλαμβάνω πως υπάρχουν ζητήματα εμπιστευτικότητας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ε, thank you that... Ευχαριστούμε. Με ενημερώνουν ότι το κείμενο έχει γίνει διαθέσιμο για τους κοιόδες, χωρίς καμία εξαίρεση. Δικό μου λάθος, συγγνώμη. Επόμενος ομιλητής, ε, έχω εδώ τη λίστα των μελών της ε, ομάδας μελέτης και παρακολούθησης, Μαρτίν Σάκε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Γενικά είμαι ικανοποιημένη με το σχέδιο ψηφίσματος. Πιστεύω ότι καλό είναι να μην είναι πολύ μεγάλο και θα επανέλθω σε συγκεκριμένα σημεία για αυτό το θέμα. Επίση, χαίρομαι που τονίζουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη και όχι της Κομισιόν του Κοινοβουλίου ξεχωριστά. Είναι σημαντικό και θα Πρέπει να αντακατοπτρίζεται ο τρόπο συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και εντό του κοινοβουλίου αυτού μεταξύ επιτροπών και σε σχέση με τον εμπορικό τομέα αλλά και με την κοινωνία των πολιτών και το κοινό. Θα το τονίσω πολλέ φορέ ότι η δημόσια στήριξη είναι ουσιαστική για αυτή τη διαδικασία ώστε να έχει επιτυχία έκβαση. Χαίρομαι λοιπόν που θα γίνει αυτή η ακρόαση σε αυτή την Επιτροπή και θα κάνω και κάποιες προτάσεις και ομιλητές ώστε να είναι πιο ελκυστική ακροσία για το κοινό. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να έχουμε κάποιο shopping list, δηλαδή εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύση. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί κομμάτι τη εντολής και χαίρομαι που τώρα συμπεριλαμβάνεται η ισχυρή ε, προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων. Ε, μάλλον δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται αυτό, γιατί αν περιλαμβάνεται αυτό, τότε θα περιλαμβάνει ο καθένα τις δικέ του επιθυμίες και στο σημείο 14 πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συμπεριλάβουμε σε αυτό το πλαίσιο για λόγους ε, προκλήσεων όπως τις βλέπει το κοινό. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς. Μάθαμε ότι ήταν ένα μάθημα από την απώλεια διαφάνειας ε, στο παρελθόν και πως ε, δυσχεραίνει τις διαδικασίες εμπορικών συμφωνιών. Θα πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε την ανάγκη για διαφάνεια. Δύο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, επίσης ε, και όσον αφορά την εντόλη, αλλά και πιο συγκεκριμένα για την πρόοδο, για την εξέλιξη της απαγόρευσης, ε, της άρσης της απαγόρευσης για το βόλιο κρέος και πώς αντιμετωπίζουμε τα κανονιστικά εμπόδια θα αντιμετωπιστούν συνολικά ή ξεχωριστά. Είναι σημαντικό ερώτημα αυτό, σχετίζεται με πολλά αρχεία και θα ήθελα πολλούς φακέλους και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις γι' αυτό. Εκτός αυτού θα ήθελα να σας ρωτήσω για το, την αύξηση των υπηρεσιών, γιατί η μελέτη της Επιτροπής εστιάζεται στα αγαθά, ενώ η υπηρεσία ουσιαστικά είναι η πλειοψηφία των εμπορικών συναλλαγών μας. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψη σας γι' αυτό. Κλείνω εδώ, ώστε οι υπόλοιποι συνάδελφοι να προλάβουν να παρέμβουν και αυτοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην ε, σύνταξη αυτού του σχεδίου ψηφίσματος. Έχω λάβει υπόψη πολλά από τα σχόλιά σας και φυσικά θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μελέτης ώστε να βελτιώσουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Ο Ρόμπερτ Θέρντι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε ίσως να κόψουμε μερικά πράγματα από αυτό το έγγραφο, αλλά σε γενικές γραμμές ε, είναι εξαιρετική η δουλειά που έχετε κάνει. Για να επιστρέψω όσο είπε μόλις η κυρία Σάκο, αναφέρατε την κατάσταση για το βόλιο κρέα. Υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος εδώ και το λέω επανειλημμένος. Η Γεωργία να παρέμβει σε αυτό, σε αυτή την πραγματική ευκαιρία για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μεγάλο εμπορικό μπλοκ με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αποτελεί τεράστια ευκαιρία και για τους δυο μας να αποτελέσουμε σημαντικό παίκτη παγκοσμίω. Και δεν λέω ότι η Γεωργία απαραίτητα θα Μπορεί, μπορεί να το καταστρέψει ουσιαστικά, γιατί η Γεωργία πάντα έχει ρευστότητα. Συναντήθηκα χθε με τους Καναδούς για να συζητήσουμε τη συμφωνία με τον Καναδά. Και σε κάθε περίπτωση φαίνεται όλοι να ανησυχούν για τη γεωργία. Αλλά ουσιαστικά όταν καθόμαστε και συζητάμε τις λεπτομέρειες γύρω από ένα τραπέζι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Είναι αρκετά εύκολα τα θέματα. Τώρα όσον αφορά το βόλιο κρέας δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει τους Ευρωπαίους αγρότες. Και ξέρω ότι ειδικότερα οι Γάλλοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο πρόβλημα ότι ε, τρέφουν τα ζώα τους οι Αμερικανοί με γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν είναι αποδεκτό και μιλάμε για 150 ευρώ κατά τόνο διαφορά στη τιμή. Συνεπώ βρίσκονται σε μειονεκτική θέση οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που αγοράζουν αυτές τις ζωοτροφές που δεν είναι γενετικά μεταλλαγμένες. Αποτελεί τεράστια ευκαιρία. Χαίρομαι που παίζει ρόλο το κοινοβούλιο σε αυτό. Την περασμένη εβδομάδα κάνατε την δήλωση τύπου στο Στρασβούργο και κάποιος ρώτησε τι θα κάνετε για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπε θα σας κρατήσω ενήμερους. Πρέ, πιστεύω πρέπει να είμαστε πολύ ενημερωμένοι και να παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις και ελπίζω κύριε Πρόεδρε να με σε αυτό. Πιστεύω ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Yes, yes, thank you. Definitely, I think that... Uh, Ευχαριστώ. Νομίζω πως οπωσδήποτε θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες ενημέρωσης από τις διαπραγματεύσεις και αυτό είχα τονίσει ε, σε κάποιο σχολείο μου πως πρέπει να ενημερωνόμαστε από την Κομισιόν πριν και μετά από κάθε διαπραγμάτευση. Έτσι αυτά για να απαντήσω στις αντιδράσεις του Επιτρόπου Ντεχούχτ όταν ήρθε και μας είπε πως θα ενημερώσει το Κοινοβουλίο. Δεν μας αρκεί αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να πούμε πριν και μετά από κάθε γύρο για να παρακολουθούμε βήμα-βήμα τις διαπραγματεύσεις και να έχουμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε και τις δικές μας θέσεις. Γιατί αυτοί θα διαπραγματευτούν, θα αποφασίσουν, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις μας, βήμα-βήμα, γύρω-γύρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, όπως είπε και η και υπάρχει τώρα η μελέτη που είχαμε αναθέσει στο London School of Economics. Πολύ σημαντική μελέτη για τον οικονομικό αντίκτυπο της συμφωνίας και τα διάφορα επίπεδα φιλοδοξίας. Στο πιο ε, υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας, όπως είπα. Πρέπει να διαβάσουν όλοι τη μελέτη. Έγινε μια παρουσίαση χτες από την Κομισιόν σε κάποιους ε, συμβούλους ε, και βοηθούς βουλευτών της Επιτροπής και νομίζω πως η μελέτη αυτή πρέπει να μελετηθεί. Γιατί βεβαίως ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το επίπεδο της ανάλυσης και ο βαθμός της ανάλυσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο Στέρντο ότι μπορούμε και στην Ευρώπη να εισάγουμε σόγια ε, μεταλλαγμένη. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Κάποιοι θέλησαν να κάνουν και σόγια στην Ευρώπη χωρίς να ε, περιέχει μεταλλαγμένα προϊόντα, αλλά ο καθένας μπορεί να τα Είπαμε και αυτό είναι το σλόγγαν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα κάνουμε την ε, ευρύτερη οικονομική ζώνη στον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρώπη το κάνει αυτό και από τη στιγμή που έχουμε αυτή την φιλοδοξία θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας και τα κατάλληλα μέσα που θα μας επιτρέπουν να κάνουμε και αξιολόγηση του αντικτύπου, των επιπτώσεων. Είπατε ότι θα υπάρχει μία μελέτη, αλλά θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα όλων των προηγούμενων μελετών και κάθε φορά που τελικά γίνεται μία ε, μελέτη ε, πριν από μία συμφωνία, δίδονται πολλές υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται εκ των υστέρων. Εάν λοιπόν, όπως λέγεται, αυτή η συμφωνία θα είναι η πιο σημαντική, θα πρέπει και εμείς τη μεθοδολογικά μέσα που διαθέτουμε να τα προσαρμόσουμε πριν από τη διαπραγμάτευση και όχι απλώς και μόνο μετά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι σκανδαλώδε. το ότι σε ένα κείμενο προς το Συμβούλιο Επιτροπή λέγει ότι αν υπογράψουμε όλες τις συμφωνίες ε, ελεύθερων συναλλαγών θα έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 2%. Ποιο μπορεί να το λέει κάτι τέτοιο. Εγώ είδα και άκουσα διάφορους οικονομολόγους για αυτό το θέμα, το μόνο που τους έκανε ήταν να γελάσουν αυτά που λέγονται. Σήμερα η κοινή γνώμη που γνωρίζει ποιες είναι οι δυσκολίες και η κρίση, τι να πει βλέποντας αυτό το χαρτάκι που λέει δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία επένδυση, να κάνουμε τίποτα στην Ευρώπη, ό,τι ανάπτυξη ε, θέλουμε με 2 εκατομμύρια θέσει απασχόληση θα το επιτύχουμε υπογράφοντα μια τέτοια συμφωνία. Όταν δίδονται τέτοιε υποσχέσει, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί διότι δεν μπορεί να ψεύδεται με τέτοιο τρόπο ένα θεσμικό ευρωπαϊκό όργανο. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν να είναι πάρα πολύ πιο αυστηρό και να κάνει την σωστή αξιολόγηση για μια τέτοιο είδους συμφωνία. Η απελευθέρωση και στις πολιτικές μας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια πραγματικά έλαβε τη μερίδα του λέοντος και ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα σήμερα. είμαστε πιο σοβαροί. Η πρώτη μου παρατηρήση ήταν αυτή. Η δεύτερη. Αυτή η διαπραγμάτευση όπως ελέγχθη δεν είναι μια διαπραγμάτευση ή περιθωριακά μια διαπραγμάτευση που αφορά τα τελωνιακά ε, τέλη. Θα συζητήσουμε προδιαγραφές, κανόνες, κανονισμούς. Και όταν μιλούμε για τέτοιου είδους προβλήματα, τι κάνουμε. Κάνουμε μία επιλογή από τις κοινωνίες μας, τις δημοκρατικές, είτε αφορώνται οι δημόσιες υπηρεσίες, η ευημερία των ε, ζώων, τα πνευματικά δικαιώματα, κανόνες επίπεδου. Πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά όλες τις κοινωνίες μας στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια πρωτίστως πολιτική συμφωνία και δευτερευόντως εμπορική. Το να μην μπορούμε να ξέρουμε σήμερα οι πολίτες της Ευρώπης βάσει ε, ποιων στοιχείων θα διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου φαίνεται ότι είναι παράλογο ακόμη και στην παρούσα κατάσταση της Ευρώπης σήμερα. Υπάρχει δυσπιστία προς την Ευρώπη εκ μέρους των πολιτών της Ευρώπης και εξ ονόματος των πολιτών της η Ευρώπη διαπραγματεύεται για, με, κάνοντας κάποιες επιλογές στην πλάτη τους, τις οποίες δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για το τι ακριβώ θα συμβεί. Και όπως λέγεται, οι αποφάσεις που θα πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε διάφορα ψηφίσματα θα πρέπει συνοπτικά και λεκονικά τι να λένε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. βασικά συμφωνούμε με ό,τι κάνετε. Ακούστε, εάν θέλετε πραγματικά να λάβουμε σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό, θα πρέπει για κάθε σημείο της διαπραγμάτευσης να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ήδη σε μια κατάσταση ποδέστερη, αν θέλετε, σε σχέση με το Συμβούλιο και θα πρέπει για τα διάφορα σημεία αυτά να γνωμοδοτήσουμε. Τελικά, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, ακόμη μια φορά βρισκόμαστε σε μια πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη εξαιρετικά πολύπλοκη. Ζητώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντί να βιαστεί. Για αυτή τη διαπραγμάτευση να ζητήσει, να απαιτήσει, να υπάρξει χρόνος ε, μελέτης όλων των σημείων της διαπραγμάτευσης και αντί να πούμε στην Επιτροπή και να πει ο κύριο Ντεγκούχο, επίτροπο, Ω, ε, πέτυχα την καλύτερη εμπορική συμφωνία. Και χάσει αυτή τη συμφωνία ο πρόεδρο Μπαγόζο να έχει τρομερέ διεθνεί φιλοδοξίε όταν θα φύγει από την Επιτροπή, δεν μα ενδιαφέρει. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι εάν συναυτεί αυτή η εμπορία να είναι συμφωνία ποιότητε και να την αποδεχθούν και να την προωθήσουν και να την ε, υποστηρίξουν οι πολίτες της Ευρώπης και όχι να είναι το κερασάκι στην τούρτα της Κομισιόν. Συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που αναφέρετε. Στην παράγραφο 15 με την κυρία Σάκα, εκεί ακριβώς αναλύονται αυτές οι ενισχύες. Ας ακούσουμε τα λοιπά μέλη του ομάδας εργασίας των... από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αναφερθήκατε ξανά στους συνολικούς στόχους της συμφωνίας και συμφωνώ με αρκετά από τα πράγματα που ανέφερε η Γιάννη. Συμφωνώ με την προσέγγισή της και με το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πριν από την έκδοση της εντολής και να καταλήγει σε μια θέση αρχής. Και αφορμή είναι η σημερινή ε, συζήτηση. Δεν έχουμε ξεκινήσει καν ακόμα την συζήτηση αυτή και τι γίνεται. Έπρεπε να ορμήσουμε στην αίθουσα όπου γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Οπότε η πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για την εντόπιση της κρίσης δεν ε, αποδίδει αυτή τη στιγμή και οι πολίτες θα μετρήσουν οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με το εξή απλό μέτρο. Τι προσφέρει σε μένα προσωπικά. Προσφέρει μια προοπτική για μια καλύτερη δουλειά, για ένα και εισόδημα κτλ. Και από πλευρά περιβάλλοντος κτλ. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό. Ειδικά όταν μιλάμε για μελλοντικέ ε, συμφωνίες και διαπραγματευτικές συντολές για την ε, Κομισιόν και τα λοιπά. Οπότε για τα ζητήματα D, E και H πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά αν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία θέλουμε. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να πω. Κατά την άποψή μου, ναι, από τη σκοπιά των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ που έχουν τελματωθεί για την περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος αυτού, Μπορούμε βεβαίω να έχουμε διμερείς συμφωνίε που ξεπερνούν τις προδιαγραφέ του ΠΟΕ, αλλά θεωρώ πως η κατάταξη αυτών των συμφωνιών στο διεθνές ε, σύστημα ε, είναι τέτοια ώστε θα πρέπει να οδηγούν σε ένα πραγματικά ισότιμο και πολυμερές σύστημα παγκοσμίου εμπορίου. Γι' αυτό πρέπει νομίζω να αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία. Γιατί, γιατί υπάρχουν μεγάλοι φόβοι παντού και γι' αυτό θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει αυτή τη θέση αρχής για τις πολυμερείς εμπορικές ε, συμφωνίες και να τα πει αυτά τα πράγματα της Κομισιόν ως εντολή για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ε, θεωρώ επίσης πως Ίσως δεν θα μπορέσουμε να αποκλείσουμε όλες τις πτυχές που είχαμε μέχρι στιγμής, αλλά οι κοινωνικές, οι οικολογικές πτυχές, αυτές που αφορούν την απασχόληση και οι οικονομικές πτυχές, νομίζω πρέπει να αναφερθούν ξεκάθαρα ως κριτήρια για την πιθανή επιτυχή κατάληξη των συνομιλιών αυτών τότε θεωρώ και χαίρομαι που είναι εδώ πέρα ο συνάδελφος ε, Μίλαν Μόραν από την Επιτροπή Εξωτερικών πως πρέπει να δούμε τη γενικότερη κατάσταση του κόσμου σήμερα. Ταυτόχρονα η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εκτιμά την ε, διατλαντική συνεργασία. Οπότε αν μιλάμε ξεκάθαρα για μια εμπορική συμφωνία και συμφωνία ε, επενδύσεων, αντιλαμβανόμαστε πως δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε από το γενικότερο πλαίσιο και χρειαζόμαστε την κατανόηση των εταίρων μας. Αν δείτε και τη συζητήση στο Κογκρέσο, τα παρόμοια λένε και εκεί πέρα οι Αμερικανοί ομόλογοι. Και όταν μιλάμε για το ρόλο του Κοινοβουλίου, αυτό τα οποία υπόθηκαν για την διαφάνεια, για την αξιοπιστία και για το πώς αντιλαμβανόμαστε μια τέτοια συμφωνία, δεν σημαίνει πως θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εγκρίνει απλά τις συμφωνίες. Η εμπειρία μας από το SWIFT, την ACTA κτλ. λέει πως αν ε, μας παίρνουν σοβαρά, τότε, ε, αν ε, με συγχωρείτε δεν μας παίρνουν σοβαρά και δεν συμμετέχουμε στον διάλογο, θα αποτύχουν αυτές οι συμφωνίες στα μάτια της κοινή γνώμης. Εμείς εκπροσωπούμε ακριβώς αυτή την κοινή γνώμη, τους λαούς, οπότε ε, υπάρχει όπως σας είπα υπάρχουν αυτές τις προσδοκίες για διαφάνεια και στον τριμερή διάλογο πρέπει να έχουμε και την ε, κοινωνία των πολιτών και τα συνδικάτα και την Business Europe και τα εθνικά κοινοβούλια. Και εδώ πέρα έχει δίκιο η κυρία Τρούπελ που ανέφερε την διάδραση μεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού επίπεδου. Ευχαριστώ. Έχω κάποια αιτήματα από άλλους ε, βουλευτές επιτροπής μας, αλλά καλύτερο είναι να δώσω μόνο τον λόγο, πρώτα τον λόγο σε μέλη άλλων επιτροπών, ξεκινώντας από την Αμέλεια Σαρτόρη που είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας. Θέλετε το λόγο. Καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και για τη δέσμευσή σας και για το πόσο ήσασταν διαθέσιμος ε, να συμμετέχετε στην Επιτροπή ΙΤΡΕ σε αυτή την προπαρασκευαστική φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή ΙΤΡΕ αντιλαμβάνεται ότι το περιεχόμενο αυτών των διαπραγματεύσεων είναι πολύ φιλόδοξο. Εμείς ε, δεσμευόμαστε να συμμετέχουμε και να υποστηρίξουμε, να προσφέρουμε αρρωγή ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισμός των εργασιών εντός του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή, η δική μου επανειλημμένος ε, έχει επισημάνει πως η σχέση ουσιαστικά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής και της ε, Κομισιόν και του εμπορικού της Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου ε, έχουν τεράστια σημασία και πώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα συμφέροντα των βιομηχανιών στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά τα σημεία τα οποία μελετάμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι δίδεται κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν πιθανώς για το κατά πόσο θα μπορούν να συμπεριληφθούν στα θέματα που θα συζητήσουμε και εδώ. Το πρώτο σχετίζεται με την ψηφιακή ελευθερία και το cloud computing Επ' αυτού ξεκινάμε μια εργασία στην Επιτροπή Ήτρε. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το θέμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως επίσης και για το θέμα της ασφάλειας πληροφορικής. που ώστε να επιτευχθεί ο κυριαρχό ρόλος των ΗΠΑ και τη ευρωπαϊκή ε, παγκοσμίω, ε, αυτό το θέμα θα είναι πολύ σημαντικό και για εμάς. Ένα άλλο θέμα για το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να, υπάρξει, να συνεργαστούμε είναι το θέμα της ενέργειας. Αυτό είναι ένας τομέας όπου φυσικά η δική μου επιτροπή έχει αναλάβει ιδιαίτερε δεσμεύσει. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε μια έκθεση πρωτοβουλία για την ενέργεια γενικότερα, για την ενιαία αγορά, για τις νέες ευκαιρίε των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά μετά όσα νέα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο για την ενέργεια και αυτή και ανταλλαγή απόψε με τις ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα. Και πάλι θα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας, εμείς ως Επιτροπή Ήτρε, το λέω και εκ φίλων, των συναδέλφων μου, για να συνεργαστούμε για τη συνοχή των διαπραγματεύσεων που θα λάβουν χώρα και που θα πρέπει πάντα, αυτό εμείς έχουμε επισημάνει συχνά και στην Κομισιόν, πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα και τα προβλήματα της Ένωσης όταν ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε μια συμφωνία. Μερικές φορές ε, ήταν επιφανειακή λίγο η αντιμετώπιση μέρους της Κομισιόν. Γι' αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει ένα ισχυρό ρόλο του Κοινοβουλίου σε όλα τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να επιδείξουμε συνοχή μεταξύ των δράσεων εξωτερικής πολιτικής και των δράσεων εσωτερικής πολιτικής. Και φυσικά θα πρέπει να συμμετέχει και η Ήτρε στις πολιτικές με τις οποίες ασχολείται. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας και ελπίζουμε ότι θα είναι επωφελή η συνεργασία μας. Ακολουθεί Φρανσίσκο Χωσέ Μιλάν. Μον εκ ΑΦΕΤ. Έχετε το λογοπακό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ΑΦΕΤ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να συμμετάσχουμε στη συζήτηση σήμερα. Όπως ελέγχθη ήδη, πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα φέρουν μία νέα πνοή και ζωτικότητα στις σχέσεις ΕΕ. Είναι λοιπόν ιστορικής σημασίας ευκαιρία για να μπορέσουμε ε, να κάνουμε ένα νέο βήμα προς τα μπλος και να προοδεύσουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και πέραν αυτής της ε, διμερούς διαπραγμάτευσης ε, τι θα γίνει στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης για όλους. Τώρα, για να επανέλθουμε σε αυτή τη διμερή σχέση, νομίζω ότι είναι ιστορική στιγμή. Μιλούμε συνέχεια για το pivot προς την Ασία, το ρόλο της Ευρώπης από τη ΣΥΠΑ. Πιστεύω ότι ε, πολλοί πίστευαν κάποια στιγμή ότι η Ευρώπη ε, βρίσκεται σε φθήνουσα κατάσταση σχέση με τη σχέση με την ΥΠΑ σήμερα, διαψεύονται. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο, ότι θέλουμε να έχουμε και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού μία ισχυρή στέθη και συνεχίζουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία τη στιγμή αυτή την οποία αντιμετωπίζουν ε, και οικονομικά προβλήματα τόσο σημαντικά οι χώρες της δύση, όπως λέγαμε παλιά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι πολιτικό και οικονομικό σημαντικό μήνυμα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και, και θεσμικά αν θέλετε την υποχρέωση να κάνει στα πλαίσια της κοινή εξωτερικής πολιτικής και εξωτερικής εμπορικής πολιτικής τέτοιου συμφωνίες και συμφωνώ με τον Πάκο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οικονομική συμφωνία με πολιτική ε, απόχρωση, μια πολιτική συμφωνία με οικονομικές αποχρώσεις. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σάρα Λόφορντ. που είναι αυτή την προσωπία που έχει να κάνει με τις σχέσεις με το Αμερικανικό Κογκρέσο. Ας ακούσουμε λοιπόν την Σάρα, μέρος αντιπροσωπείας με τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για το πώς ε, συμπεριλαμβάνονται και τις άλλες επιτροπές στην ε, διαδικασία αυτή και τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες. Και το εκτιμώ αυτό όπως ε, και η αντιπροσωπεία μας στο σύνολό της υπό την προεδρία του κυρίου Έλερ. Νομίζω πως έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ψήφισμα και δεν θα μακρηγορήσω με βάση βέβαια τα δεδομένα του Κοινοβουλίου. Νομίζω πως αυτό το οποίο μόλις είπατε για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή του Κογκρέσου είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε είναι ιδιαίτερα σωστή η παράγραφος 18, γιατί βεβαίω υπάρχουν διαφοροί φορείς στα δύο αυτά κοινοβούλια, νομοθετικά σώματα και υπάρχει μια σειρά σχέσεων μεταξύ των τεσσάρων αυτών νομοθετικών σωμάτων και θεωρώ πως η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στον διατλαντικό νομοθετικό διάλογο θα μπορέσει πράγματι να παίξει ένα σημαντικό ρόλο εδώ πέρα και έχουμε νομίζω μια κοινή συνεδρίαση τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου οπότε και ελπίζω θα έχουμε μια συνεισφορά στη διαδικασία αυτή. Επίσης αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λένε όσοι υπενθυμίζουν στην Κομισιόν πως πρέπει να εμπλέκει στην διαδικασία το Κοινοβούλιο. Ελπίζω να έχει διδαχτεί από τις υποθέσεις SWIFT και ACTA πως δεν έχει νόημα ε, να έρχεται ε, μόνο μετά από τις διαπραγματεύσεις και να μας λέει αυτό είναι και άμα σας αρέσει. Είμαι σίγουρη πως η Κομισιόν θα θυμάται αυτές τις εμπειρίες της και δεν θα θέλει να τις επαναλάβει. και είμαι σίγουρη πως ε, εδώ πέρα μας ακούσει ο Επίτροπος κ. Δεχούχτ. Η προσωπική μου τώρα προτίμηση είναι υπέρ της συμφωνίας αυτής. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Ζαντό που λέει πως ο φιλελευθερισμός είναι η πηγή όλων των κακών. Ως φιλελεύθερη με κεφαλαίο φι θεωρώ πως ο περισσότερος φιλελευθερισμός θα κάνει καλό. Οπότε υποστηρίζω και την ιδέα πως το ελεύθερο εμπόριο ε, και οι επενδύσεις θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας ε, και την ε, ε, οικονομική ευημερία, αλλά θα πρέπει βέβαια να δούμε τις λεπτομέρειες καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Κάτι τώρα στο οποίο θα ενθάρρυνε την Κομισιόν είναι να φροντίσει πως δεν θα υπάρχουν παγίδες στους επόμενους μήνες. Προφανώς δεν είναι η ιδιωτικότητά μου τα ζητήματα αυτά, τα αριθμιστικά, αλλά η επίλη, η... τερματισμός του προγράμματος ε, γαλακτικού οξέως ε, επιλήθηκε νομίζω επιτυχώς. Και ήταν περίεργο το ότι συνεχισόταν για τόσο καιρό και αναρωτιέμαι αν υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει η Κομισιόν να τα δει ε, για να μας ε, εκθέσουν ε, κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας. Όπως είπα δεν είναι το πεδίο αρμοδιότητάς μου. Μπορούμε να δούμε το στεάρ, το ζωικό λίπος. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το οποίο λύθηκε ε, γρήγορα και δεν θα διακινδυνεύσει την προ... των διαπραγματεύσεων. Η άποψή μου, λοιπόν, και της Επιτροπής ε, ΛΥΜΕ ε, αφορά κυρίως πράγματα όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων. Μια συναρπαστική προοπτική είναι το ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο διατλαντικό, το οποίο θα μας επιτρέψει να ορίσουμε παγκόσμιες προδιαγραφές και κατά την άποψή μου αυτό είναι ε, καλύτερο από κάποιες άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε. Οπότε εντάξει θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους ε, ιτημένους ε, και χαμένους και κερδισμένους, αλλά συνολικά το αποτέλεσμα νομίζω θα είναι θετικό. Τελευταίο. Ένα τελευταίο ζήτημα. Είδα πως ε, η παράγραφος 16 λέει πως πρέπει να φροντίσουμε την ποιότητα ε, και να μην βιαστούμε. Ναι βεβαίως, αλλά να μην χρονοτριβούμε κιόλας. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, μπορεί να είμαστε και γρήγοροι και με ε, ποιότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Ας επανελθούμε στα υπόλοιπα μέλη αυτής της Επιτροπής, επειδή έχουμε λιγότερα από 15 λεπτά πριν ξεκινήσει η συνεδρία των συντονιστών, θα χρειαστεί να περιορίσω τον χρόνο των παρεμβάσεων στο εξή στα τρία λεπτά, διότι έχω πολλά αιτήματα Μπερτλάνγκε από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι το ψήφισμα αυτό αφορά την εντολή και εδώ πέρα έχει ε, η κυρία Ροβολτή και πως αυτό είναι το κέντρο αυτού του ψηφίσματος και βεβαίω υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε να πούμε πως το ότι θέλουμε να έχουμε κάποιες προδιαγραφές που θα βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικότερα στην Αμερικάνικη αγορά είναι καλό. Θέλουμε να μειώσουμε τα μη δασμολογικά εμπόδια και να διασφαλίσουμε πως θα έχουμε αεφορία και από πλευρά προστασία περιβάλλοντο, αλλά και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Βεβαίω, Αν δούμε στις, ε, τι γίνεται στη ΣΥΠΑ, ε, ξεκαθάρισαν κάποιοι γερουσιαστές πως έχουν και αυτοί κάποια συμφέροντα που είναι αντίθετα με τα δικά μας. Οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, όπως παραδείγματο χάρη το ζήτημα του ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε κρέας με ορμόνες ανεφόρων στην ευρωπαϊκή αγορά ή κρέας αποκλωνοποίηση στην ευρωπαϊκή αγορά ή ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι ε, να δεχτούμε κοτόπουλα πλημμένα με χλωρίνη στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτά είναι συμφέροντα πολύ ισχυρά στις ΗΠΑ και πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή τοποθέτηση ή το θέμα α, των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις που είναι διαφορετικές από αυτές των ΗΠΑ και τρίτον, το είπαν και οι συνάδελφοι ε, από τις άλλες επιτροπές, η προστασία των δεδομένων. Έχουμε ήδη πολύ ε, έντονες συζητήσεις για αυτό το ζήτημα. Οπότε, δεν είναι τυχαίο το ότι κάποιες αμερικανικές επιχειρήσεις ε, ε, έφεραν τους ε, σερβερ ε, στην Ευρώπη και όχι στις ΗΠΑ, γιατί ακριβώς εδώ πέρα ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οπότε ναι, διαπραγματευόμαστε, έχουμε κάποια επιθετικά συμφέροντα, αλλά έχουμε και κάποια αμυντικά, αν θέλετε, και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα στους Αμερικανούς εταίρους μας, έτσι ώστε να είναι σαφές και ποια είναι η δική μας στάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η Ελίζα Μπεθκόσιγκερ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Θεωρώ πως πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν κάποια σημαντικά ζητήματα και ακριβώς πριν αρχίσουν διαπραγματεύσεις πρέπει να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να υποστηρίξω αυτούς που ανέφεραν πως ε, υπάρχουν πολύ ευαίσθητα ζητήματα στο πλαίσιο αυτής της εμπορικής συμφωνίας και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δημόσιες συζητήσεις για αυτά τα θέματα, για τις εισαγωγές ε, γενετικά τροποποιημένων ε, οργανισμών ε, εδώ πέρα όμως θέλω να διαφωνήσω με τον κύριο Ζαντό. Δεν εισάγονται αυτά έτσι απλά στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολύ αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί. Θεωρώ λοιπόν πως αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει ανοιχτά Ακριβώς γιατί υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στους καταναλωτές για αυτά τα ζητήματα και το θέμα του κρέατος με ορμόνες ξέρουμε πως είναι ε, πολυετής διαμάχη ε, για τις ε, ΙΠΑ και καλό θα ήταν να ορίσουμε στο ψήσιμο μία βάση για την διατροφική ασφάλεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπω σημαντικό θα είναι και το θέμα των γεωγραφικών ε, ενδείξεων ε, που έχει η Ευρώπη, όπου έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παράδοση και βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ γεωγραφικής ε, προστασίας και προστασίας της Και Έχουμε, εδώ πέρα νομίζω πρέπει να έχουμε μια στεναρή θέση για να καταλήξουν επιτυχώς οι συνομιλίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αρίβεντερ. Τους σοσιαλιστές. Λοιπόν, αυτό το προσχέδιο ψηφίσματος μου φαίνεται ότι είναι αρκετά καλό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά βεβαίως είναι βελτιώσιμο όπως οποιοδήποτε σχέδιο ψηφίσματος. Και είπατε ευθύ εξ αρχής ότι αναμφίβολα πρόκειται για τη Συμφωνία Ελευθέρου Βολίου που είναι η πιο ε, σημαντική και η πιο φιλόδοξη. Και οι επιπτώσεις του βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν μη τι άλλο και για τις εμπορικές σχέσεις μας. Εάν το συνυπογράψουμε, το 60% των εμπορικών μας ε, σχέσεων θα γίνονται ε, η βάση αυτής της ε, διμερούς συμφωνίας. Τα πλαίσια λοιπόν της συστήματος του παγκοσμίου πολυμερών συμφωνιών. Ξέρουμε μια τέτοια διμερής συμφωνία τι είδους μειονεκτήματα έχει. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα ποσοστό το οποίο ε, πριν από 10 χρόνια ανεργόταν στο 25%. Άλλαξαν τα πράγματα, ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις, οι θετικές, οι αρνητικές και ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και σε κανονιστικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν, όντως, για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το ερώτημα είναι το εξή. Υπάρχουν φήμε για τι προθεσμίε. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά έχουμε σχεδόν μόνο ένα χρόνο στη θέση μα. Κάποιοι επίτρεποι αλλά και κάποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να συναυθεί κατά τη διάρκεια της δικής τους ε, θητείας η εμπορική αυτή συμφωνία. Πράγμα το οποίο δεν αντιτίθεται με αυτά που προτείνεται. ότι ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει εμφανθύνοντας το όλο θέμα και κάνοντας τα πάντα με διαφάνεια. Θα έχουμε όμως τον χρόνο να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με μεγάλη σοβαρότητα αυτή την τόσο εκτεταμένη και σημαντική συμφωνία. Διότι όντω πρόκειται για μια φιλόδοξη συμφωνία, σημαντική αλλά και πάρα πολύ πολύπλοκη. Διότι υπάρχουν πολλά σημεία σύγκλησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ στον πολυπολικό κόσμο στον οποίο ζούμε. Δεν υποτιμώ τα σημεία σύγκλησης, αλλά υπάρχουν και πολλά σημεία αποκλήσεων, δύσκολα σημεία που αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες. Το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η πολιτιστική εξαίρεση, αυτή που αφορά τα οπτικοακουστικά μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα, η προστασία των καταναλωτών σύμφωνα με τις δικές αντιλήψεις, ε, τα κλιματικά προβλήματα, η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι λεπτομέρειες αυτά ή δευτερεύουσα σημασία θέματα. Θέλουμε να μπορέσουμε να επιδείξουμε αυτή τη συμφωνία, αλλά όχι με οποιαδήποτε τίμημα. Ευχαριστώ. Έχουν κλείσει αιτήσει ε, για να λάβετε το λόγο. Ο τελευταίο ομιλητή είναι ο Ντανιέλ Κασπάρη. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το σχέδιο ψηφίσματος γιατί δεν συμπεριλάβατε όλα τα προβλήματα που συζητάμε εδώ και χρόνια στο Κοινοβούλιο, αλλά πάρα πολύ ε, συνετά ε, επιλέξατε κάποιες έξυπνες διατυπώσεις. Θέλω πραγματικά να ζητήσω στους να σκεφτούν το τι πρέπει να μπει σε αυτό το ψήφισμα. Δεν έχουμε κάποια διαφωνία στα διάφορα προβλήματα. Υπάρχει όμως σαφή, σαφής ε, τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κρέας με ορμόνες. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα πολλές φορές, έχει τοποθετηθεί πολλές φορές και έχουμε μια συνένεση. Θεωρώ πως η Αμερικανική πλευρά γνωρίζει εξίσου καλά με εμάς τα προβλήματα, το θέμα ε, των σπόρων, πολιτιστικών αγαθών κτλ. Το να, το, ξαναγρά... το να μην γράψουμε κάτι δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά ε, πρέπει να το γράψουμε εδώ πέρα. Γιατί, γιατί πρώτον η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής για όλα αυτά τα ζητήματα και δεύτερον γιατί ε, ξαφνικά όλα τα υπόλοιπα ζητήματα θα έχουν πολύ λιγότερη σημασία. Δηλαδή θα έχουμε 5-10 ζητήματα, αλλά άλλα που είναι εξ, εξίσου σημαντικά, π.χ. Ε, προδιαγραφές ε, της βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν θα τα αναφέρουμε. Οπότε τι θα λέμε ως Κοινοβούλιο, πως ε, αυτά που αναφέρουμε είναι πολύ σημαντικότερα, αυτά που δεν αναφέρουμε είναι δευτερεύοντα. Και ότι δεν στηρίζουμε την Κομισιόν στα υπόλοιπα. Γι' αυτό παρακαλώ όλους συναδέλφους να σκεφτούν το τι θέλουμε να μπει σε αυτό το ψήφισμα. Καλό είναι λοιπόν να μην αναφερθούν αυτά τα πράγματα ρητός και η θέση του Κοινοβουλίου σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι, όπως είπα, ούτως ή άλλως γνωστή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Έχουν ήδη υποθεί πολλά. Και αυτά που είπε ο κύριος Κασπάρη μόλις, ε, ότι αυτό είναι το ψήφισμα, πρέπει να το προσαρμόσουμε έτσι όπως είναι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παρακολουθούμε όμως κάποια πράγματα και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό να συνεχιστούν οι διάλογοι και οι συζητήσει με την Κομισιόν για τα ζητήματα όπως αυτά που αναφέρθηκαν. Ακούσαμε για τις ορμόνες στο βόλιο πολλά από τα γεωργικά προϊόντα μας απασχολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σκέφτηκα και κάτι άλλο, ότι έχουμε κι άλλο ένα θέμα με αυτή τη συμφωνία. Αυτή τη στιγμή συνάπτουμε τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με τον Καναδά. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ξεκινάμε μια άλλη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με εμπορικά μπλοκ που έχουν μεταξύ τους ε, ήδη κάποιες εμπορικές ε, διευθετήσεις. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Μπορεί να διαπραγματευτούμε ένα πράγμα με τον Καναδά και κάτι άλλο με τις ΗΠΑ και αυτό να έρθει να, δημιουργήσει, να έρθει σε με τις συμφωνίες μεταξύ τους. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να το παρακολουθούμε. Και να τα λαμβάνουμε υπόψη στη συνεργασία μας με τις Κομισιόν, να φροντίσουμε, όπως είπε προηγουμένως η Σάρα, να μην ε, δημιουργηθούν ε, παγίδες. Αυτού του είδους τα πράγματα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να παρακολουθούμε. Τώρα για αυτό εδώ το ψήφισμα εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τα όσα έχουμε εδώ σε αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίτια ε, Σάκα. Ε, μου είπαν ότι θέλετε να μιλήσετε. 15 δευτερόλεπτα. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Ξέχασα κατά την πρώτη μου παρέμβαση να ρωτήσω κατά πόσο έχετε σκεφτεί ή κατά πόσο θα έπρεπε να σκεφτούμε, μπορούμε να σκεφτούμε το ρόλο της Τουρκίας σε αυτή τη συμφωνία, διότι είναι μέλος της Τελωνιακής Ένωσης. Πιστεύω ότι πρέπει να εκτιμήσουμε το αντίκτυπο για ένα τόσο σημαντικό οικονομικό εταίρο. Σας ρωτώ λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε επικοδομητικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε την Κομισιόν πέραν των σχολείων τους για το σχέδιο ψηφίσματος, θέλουμε να μας μιλήσουν για τα εξής. Τρία. Πρώτον, υπάρχουν προηγούμενες ή παράλληλες συμφωνίες ε, για κάποια ευαίσθητα ζητήματα, όπως τις εξαγωγές βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αυτό που ανέφερε η Σάρα Λόφορντ ή ε, άλλα ζητήματα που ίσως να γνωρίζει η Κομισιόν καλύτερα από μένα. Δεύτερον, το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Ποια είναι η άποψη της Κομισιόν για το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Τρίτον, Τουρκία. Ευαίσθητο θέμα. Και πιστεύω πολύ σωστά το ανέφερε η Μαρία Σάκη. Έχετε το λόγο λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ντέμιαν Λέβη, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα το πρωί, ζητώ συγγνώμη, πέντε λεπτά. Πιστεύω θα είμαι συντομότερο και από πέντε λεπτά. Πρώτα απ' όλα συμφωνούμε με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Ζαν Ντεματία θα είναι εδώ αύριο στην ε, συνάντηση κλεισμένη των θύρων. Πολλά έγκυρα σημεία αναφέρθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση από μέλη της ΣΥΝΤΑ όπως και των άλλων επιτροπών που έχετε καλέσει, ΑΦΕΤ, ΙΤΡΕ και της αντιπροσωπείας ε, για τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Δεν ήρθα εδώ για να σας πω τι πρέπει να συμπεριλάβετε και τι όχι στο ψηφισμά σας. Όπως λέμε στα γαλλικά, το να ράβεις και να ξεράβεις είναι πάντα δουλειά. Προσωπικά μου αρέσει πολύ ο μινιμαλισμός, ε, ότι less is more, όπως λέμε, ειδικότερα μετά τις αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διάφορες συνθήκες στις οποίες συμμετείχαν οι Ευρωπα... συμφωνούν οι ΕΠΑ γενικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς ε, θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι άδικο να επικρίνουμε τα όσα είπε η Κομισιόν Στρασβούργο. Αλλά είχε αναλάβει και δύο δεσμεύσεις και πολλές δεσμεύσεις όπως θα θυμάστε για να ενημερώνει το κοινοβούλιο, να αναμένει τα ψηφίσματά σας πριν περάσουμε σε προσωρινή εφαρμογή και έχει δείξει ο Επιτροπό δέσμευσή του στην Επιτροπή ΙΝΤΑ και στο Κοινοβούλιο γενικότερα. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν ζητάτε να ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, διότι όπω καταλαβαίνετε πρέπει και εμεί να κάνουμε τη δική μα δουλειά, να διαπραγματευτούμε τη συμφωνία. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τι τρει ερωτήσει σα. Υπάρχει μια παραγραφό στην τελευταία έκθεση αυτή τη ομάδα υψηλού επίπεδου για την ανάπτυξη και τη εργασία. Εγώ ε, προέδρευσα μαζί με τον Κάρλ Ντεκούχτ. Μιλήσαμε για τα ζητήματα SPS, όπου σημειώθηκε πρόοδο σε διάφορα σημείο όπως το γαλακτικό οξύ που αναφέρθηκε αλλά και άλλα θέματα έχουν ληφθεί διάφορες αποφάσεις για διευκόλυνση των εξαγωγών των προϊόντων κρέατος των αβοκάντο προς κάποια κρατημέλη και από κάποια κρατημέλη και αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ε, συμπεριλαμβάνουμε και το στέατο στέατος ε, ε, από πλευράς μας και φυσικά και το θέμα των εξαγωγών βόηου κρέατος που έχει απαγορευτεί εδώ και πολύ καιρό όπως γνωρίζουμε όλοι. Τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ακούσαμε τον πρόεδρο Μπαρούσο και τον Επίτροπο επί του θέματος πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα αλλά θα δώσουμε προτεραιότητα στην ουσία και όχι στο χρόνο ε, αλλά μετά από ξέρετε, τη διαπραγμάτευση χρειαζόμαστε και την εξέταση από υπηρεσίας, υπηρεσία, την μετάφραση και τις διαδικασίες επικύρωση. Όλα αυτά χρειάζονται κάποιο χρόνο. Και τέλος, ε, δεν πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ πριν το τέλος του παρόντος κοινοβουλίου. Δεν πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό δεδομένων όλων των βημάτων που χρειάζονται. Τέλος, όσον την Τουρκία, πολύ σωστά το θέσατε αυτό το θέμα. Έχουμε μια συμφωνία σύνδεσης με την Τουρκία και έχουμε και κάποιες δεσμεύσεις με τους ε, εταίρους μας. Ε, πρέπει να τους ζητήσουμε να ξεκινήσουν και διαπραγματεύσει με την Τουρκία, διότι θα έχουμε πρόβλημα ε, αγαθών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά δεν μπορούν να περάσουν στην Τουρκία εμέσως. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτό το θέμα της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Φυσικά εκτιμώ ιδιαίτερα την ευρεία και γενική υποστήριξη για το σχέδιό μου, αλλά όπως υπόθηκε μπορεί να βελτιωθεί και πρέπει να βελτιωθεί. Θα αναμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, άκουσα προσεκτικά τις παρατηρήσεις σας και τις επιφυλάξεις που ακούστηκαν επίσης. Πιστεύω ότι το ζήτημα κλειδί είναι ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογής του ψηφίσματος Άλλοι ζήτησαν μικρότερο ψήφισμα, άλλοι μεγαλύτερο. Ουσιαστικά για το πόσο μεγάλο θα αυτό το ψήφισμα και πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λεπτομερώς όλα τα θέματα. Θα πρέπει να αναφερθούμε στις γνωστές θέσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά κάποια ευαίσθητα θέματα. Δεν χρειάζεται να επιμείνουμε λεπτομερώς σε αυτά. Ανυπομονώ λοιπόν να λάβω τα παρατηρήσει σα, που για όσου από εσά να μου τι στείλετε εγγράφο. Και τελικά, φυσικά, θα συζητήσουμε. Θα συζητήσω μαζί σα, ώστε το σχέδιο αυτοψηφίσματο να βελτιστοποιηθεί στο μέγιστο. Τώρα, όσον αφορά τα διαδικαστικά, τη διαδικασία εμπλοκή αυτής της επιτροπή ε, με την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα τα σχόλιά μου όσον αφορά τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, ε, υπονοούν οποιαδήποτε κριτική προς προηγούμενα, προηγούμενες σχέσεις με την Κομισιόν που ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής υπήρξαν ιδιαίτερα ικανοποιητικέ. Το έχω πει επανειλημμένως. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Επίτροπος Δεκούχτ αντιμετωπίζει τη συνεργασία του με αυτήν εδώ την Επιτροπή. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτής της συμφωνίας μας ε, επιβάλλει μια διαφορετική τύπου εμπλοκή. Πρέπει να δούμε τι σκοπεύει, ποιες είναι οι προθέσεις της Επιτροπής για αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει ισότιμα στις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό το λόγο επέμεινα να συμπεριληφθεί αυτό το κείμενο ότι πρέπει να ενημερωθούμε πριν και μετά το γύρο διαπραγματεύσεων όπως γνωρίζετε. Εγώ είμαι υπέρ της, ε, του επιμερισμού των εξουσιών. Δεν θέλω το κοινοβούλιο αυτό να παρέμβει στις διαπραγματεύσεις ή να συμμετέχει, αλλά θέλω το κοινοβούλιο αυτό να γνωστοποιήσει τις απόψεις του στην Κομισιόν πριν από οποιονδήποτε γύρο διαπραγματεύσεων και να ενημερωθεί για την έκβαση κάθε γύρου διαπραγματεύσεων. Αυτό υποστηρίζω και αυτό πιστεύω η παρούσα Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίζουν. Να μην υπάρξει λοιπόν καμία παρανόηση. Αυτή είναι η γραμμή που θέλουμε. Θέλουμε απλά να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε την καλή σχέση που είχαμε με την Κομισιόν και τον Επίτροπο Ντεχούκτ και τις γενικέ διευθύνσει, τις διευθύνσει μάλλον τη Γενική Διευθύνση Εμπορίου. Και πιστεύω ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Α συνεχίσουμε λοιπόν και με τον ίδιο τρόπο σε αυτό το ζήτημα κλειδί. Ας δούμε τις άλλες προτάσεις που ακούσαμε. Ακούσαμε προτάσεις για τακτική ανταλλαγή απόψεων, ενδεχομένω μετά από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων. Μπορούμε να το εξετάσουμε αργότερα. Πριν λάβουμε κάποια θέση εδώ στην Ολομέλεια της Επιτροπής, ας λάβουμε ε, υπόψη και ας μελετήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα στην μόνιμη ομάδα για τις ΗΠΑ. Αλλά εγώ θα λάβω υπόψη όλες τις συστάσεις και προτάσεις, θα τις εξετάσουμε με σοβαρότητα και εν το χρόνο θα έρθουμε σε αυτήν την Επιτροπή ώστε να υιοθετήσουμε έναν οδικό χάρτη για τη συμμετοχή μας ε, όχι μόνο σε εργασίες της Επιτροπής αλλά και με τις άλλες Επιτροπές ε, εδώ του Κοινοβουλίου που θα συμμετέχουν σε αυτή μας την προσπάθεια με συνοχή. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 8 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το δημόσιο κομμάτι αυτής της συνεδρίασης. Καλό λοιπόν όσους δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στην συνεδρίαση συντονιστών να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Παρακαλώ το ταχύτερο δυνατόν και όσο το δυνατόν πιο ήσυχα και αθόρυβα.